Liebe Kollegin, Αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας και γι' αυτό παρακαλώ να καθίσετε κατά τρόπον ώστε να ε, μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη δουλειά μας και ό,τι ε, άλλα θέματα προσωπικά έχετε παρακαλώ να τα διακόψετε. Ξεκινάμε λοιπόν με το σημείο 13 που είναι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σχετικά με την πολιτική αναπτυξιακή ε, συνοχής για το 2011 και η, η για αυτή την ε, γνωμοδότηση είναι η κυρία Έρνα Κοστέλο, στην οποία δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είμαι σχετικά νέα Ευρωβουλευτής και πρώτη για την πρώτη μου γνωμοδότηση, ξέρετε. Οπότε, με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τη γραμματεία της Επιτροπής μας για τη βοήθειά τους και τους προσωπικούς μου συνεργάτες για την βοήθειά τους. Το 2005 αυτό σωστή συνένεση για την συνοχή για την ανάπτυξη Οπότε αυτό απαιτέλεσε μια υποχρέωση για όλες τις πολιτικές. Όλες, να έχουμε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους στόχους της ε, ανάπτυξης και έτσι αναγνωρίζεται ότι η αναπτυξιακή συνεργασία δεν καλύπτει από μόνη της τις ανάγκες των χωρών αυτών και έχουμε επομένως ε, για αυτή την συνεργασία την νομική βάση που την ενίσχυσε η Συνθήκη Λισαβόνας και το Δεκέμβριο του 2009 και έχουμε το 2008 όπου ορίζει ότι θα πρέπει η Ένωση να λάβει υπόψη τους στόχους της συνοδοσιακής συνεργασίας για τις πολιτικές σε σχέση με τις αντισώμενες χώρες. Και έχουμε επομένω την κοινωνική ρήτρα του αρθρού 9 σε σχέση με την συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επομένω έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να λάβει υπόψη τα όσα απαιτούνται για να γίνει κάτι για την υψηλή ανεργία και την καταπολέμηση της, του γενικού αποκλεισμού, την κατάρτιση και την προστασία της ε, υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός αυτής. Η η... Το σχέδιο αυτής της εκθεσής μου τονίζει το ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές διατάξεις των εμπορικών συμφωνιών. Ε, αυτές να τηρούνται και να εποπτεύεται η εφαρμογή τους. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να, ε, να, να, να έχει εδώ κάποιες δεσμευτικές διατάξεις για την απασχόληση ιδίω των γυναικών και των νέων. Και κατοχυρώνεται η ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των εργαζομένων, κοινωνική υπευθυνότητα και τονίζει το ότι θα πρέπει να έχουμε ε, την συνεκτική αναπτυξιακή πολιτική PCD. Και θα πρέπει να και κάποια ζητήματα όπως τα εμβάζουν των εργαζομένων και επίσης ε, χρήση των κοινωνικών πόρων που να καταπονημούν τον κοινωνικό αποκλεισμό, κάτι το οποίο δεν θεωρείται, δεν θεωρείται αρμοδιότητα των, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά όσον αφορά την κοινωνική πολιτική και την απασχόληση. Λέω τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβουν υπόψη περισσότερο την ένταξη των μεταναστών στη χώρα υποδοχή και αναφέρεται πιο συγκεκριμένα στο θέμα των δικαιωμάτων των μεταναστών. Και είπαμε ότι θα πρέπει να τηρηθούν αυτά τα κοινωνικά πρότυπα και εκτός των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπαμε επίσης ότι χρειάζεται μια γνωμοδότηση από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων που θα είναι το πιο σωστό να λάβει υπόψη το πλαίσιο όλων των ρυθμίσεων. Αυτό το λαμβάνει υπόψη το ψήφισμα, οπότε και θα πρέπει η Επιτροπή και το Συμβούλιο να δεσμευτούν περισσότερο όσον αφορά την ε, πολιτική της συνοχής για την ανάπτυξη. PCD. Σε σχέση με τις αντισώμενες χώρες θα μπορούσαμε όλα αυτά αντί να τα αναλάβει σε χωστή έκθεση η Επιτροπή να τα εντάξουμε στο κείμενο με τροπολογίες. Επομένως, σύντομη η έκθεση και καλοδεχούμενα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε και ε, μπορεί να είμαστε λίγοι εδώ, αλλά σε συνεργασία με τους συναδέλφους είμαι βέβαιη ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε ε, σε μία σωστή γνωμοδότηση. Τον ε, λόγο δίνω πρώτα στον κύριο Ρολό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να πω στην εισηγήτριά τη ότι για την πρώτη αυτή τη γνωμοδότηση δεν θα έχει προβλήματα ιδιαίτερα με εμά. Θα υποβάλουμε τροπολογίε και θα βρούμε σημεία σύγκληση. Παραδοσιακά η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν παρέχει αναπτυξιακή βοήθεια το πράττει σε ε, μέρη όπου υπάρχει κάποιο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεμελιώδης. Ε, αυτό είναι ένα τρόπο με τον οποίο εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε και να προωθήσουμε την κοινωνική πρόοδο και τις κοινωνικές μα αξίες και όλη την προβληματική την οποία διαρκώς επεξεργαζόμαστε εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά φυσικά μπορούν να μεταφερθούν στις ε, υποανάπτυξη χώρε, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Φυσικά τα κοινωνικά κριτήρια και πρότυπα είναι σημαντικά ζητήματα για τα οποία έχουμε μιλήσει τις τελευταίες μέρες ε, με την εκθέση της κυρίας Στανουέη και η κοινωνική ευθύνη επίσης και όλοι η πολιτική που προσπαθούμε να διεξάγουμε σε αυτόν τον τομέα. Εγώ είμαι και εκπρόσωπος του ΕΛΚ για μια πρωτοβουλία που θα μετατρέψει το 2015 σε Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, της επερχόμενης πρωτοβουλίας, θα υποστηρίξω τους προσανατολισμούς που μόλις ανέφερε η συγγήτρια, στην οποία θα στείλουμε αρκετά σύντομα τα τροπολογίες μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπουλόν. Δεν βλέπω κανένα άλλο να ζητά το λόγο τώρα. Κοιτώ και γύρω γύρω μήπως κάτι μου έχει διαφύγει. Όχι, δεν βλέπω κανέναν. Οπότε έχουμε όμως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και συγκεκριμένα την κυρία Ντομπιέσοβα που θα ήθελα πρώτα να σας δώσω το λόγο και μετά θα τον δώσω πάλι στον εισηγητή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να εκφράσω την ευχαριστησή μου για τις πολύ ωφέλιμες προτάσεις, ε, τις σημειώνουμε και θα θέλαμε και μεγαλύτερη ανάλυση ορισμένων αυτών των σημείων, των εστιακών σημείων για την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, εξερευνούμε αυτή τη στιγμή το πώς θα μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε στον διάλογο με τις δημόσιες αρχές περισσότερα θέματα συνοχής για την αναπτυξιακή πολιτική, PCD, και να χρησιμοποιήσουμε τις αντιπροσωπές μας ως κόμβους για την συλλογή σχολείων για το PCD και για κοινωνικά θέματα. Θα πρέπει να τους παρέχουμε περισσότερους πόρους και να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες για το ζήτημα, για το θεματολόγιο, ώστε να μπορέσουν να μας αποστελούν αυτοί περισσότερες ε, πληροφορίες για τις επιπτώσεις της άλλες χώρες όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου της προτινόμενης νομοθεσίας σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη από το 2009 στις οδηγίες της Κομισιόν για την εκτίμηση αντικτύπου υπάρχει απέτηση εξέτασης του αντικτύπου σε τρίτες χώρες ε, και φυσικά αυτό συμπεριλαμβάνει και τις κοινωνικές πτυχές. Ε, έχουν γίνει εκτιμήσεις από το 2009 αλλά δεν έχει δοθεί ιδέωσα προσοχή ε, για πολλούς λόγους. Ο κύριος λόγος είναι ότι βασίζονταν στις παλιές κατευθυντήριες γραμμές αλλά ε, προβλέπουμε μεγαλύτερη εξέλιξη σε αυτό το μέτωπο στο άμεσο μέλλον. Επίσης υπάρχει ένα επιπλέον σημείο αφορά το διάλογα με συνδικάτα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια από τις προτάσεις στο θεματολόγιο αυξάνει το διάλογο βασιχωρών ε, με την κοινωνία των πολιτών της κάθε χώρας ε, συμπεριλαμβανομένων των συνδικάτων. Ελπίζω αυτό να απαντά σε ορισμένα από τα σημεία, της, από τα σημεία σας. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα δίνω και πάλι το λόγο στην ε, εισηγήτρια κυρία Κοστέλο. Ε, ε, Ευχαριστώ. Όπως ε, ανέφερα, ήταν η πρώτη ευκαιρία που είχα να καταρτήσω μία έκθεση και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η εμπειρία. Ευχαριστώ και για τις προτάσεις και για την στήριξη και ε, ευχαρίστως ε, θα συνεργαστώ και με όποιον θέλει ε, κάτι παραπάνω ή να συζητήσουμε ώσπου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρξουν τροπολογίες και αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια μικρή γνωμοδότηση η οποία όμως είναι πολύ σημαντική ιδίως για την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης και γι' αυτό χαίρομαι που είχα την ευκαιρία και είμαι γνώμων που είχα την ευκαιρία να βοηθήσω σε αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει αυτά να τα εξετάσουμε εδώ ε, όπως είπατε και για τους σκιώδεις είναι σημαντικό η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 25 Ιουνίου, δηλαδή τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι και οι τροπολογίες σας παρακαλώ να ε, διατυπωθούν αγγλικά διότι δεν έχουμε την ε, δυνατότητα δυνατότητα να έχουμε εγκαίρως μεταφράσεις αν θέλουμε εγκαίρως να την ξαναδούμε στην Επιτροπή η οποία είναι υπεύθυνη για την έκθεση επί της ουσίας δηλαδή, ε, κατά τρόπον ώστε να τις ξαναδούμε και να τις προωθήσουμε. Και έτσι κλείνω αυτό το θέμα και έτσι τώρα επανερχόμαστε στο προηγούμενο σημείο, δηλαδή το σημείο 12 της ημερησίας διατάξεως και ξεκινάμε τη δημόσια κρόασή μας, μάλλον τη συνεχίζουμε. Δηλαδή, αν κάνετε μερικές σελίδες πίσω, θα δείτε ότι δίνουμε το λόγο στην κυρία Μπάστος, η οποία είναι η συγγήτρια της Επιτροπής επί του θέματος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω επίσης όλους όσους ήρθαν να μας ακούσουν σε αυτήν εδώ την ε, ακρόαση για το, τα ασφαλιστικά στην ε, Ευρώπη και, και το Ταμείο Έλληνα Οπότε και θα πρέπει να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την ακρόαση. Μιλούμε για την ε, αλληλασφάλιση που είναι μια ιστορία παλιά εις τις περισσότερες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ορισμένες πάντως ε, δεν υπάρχουν. Σε Κύπρο Τσεχία, Εστονία, Λιθουανία και Σλοβακία. Δεν έχουμε ταμεία αλληλασφάλισης. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει κοινωτική νομοθεσία για τα ταμεία αυτά. Όμως αυτά τα ταμεία αλληλασφάλισης πρέπει να υποστούν κάποια ευρωπαϊκή εναρμόνιση. Και οι χώρες οι οποίες σήμερα έχουν τη σχετική εμπειρία και εδώ και αιώνες να μπορούν να μοιραστούν και με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη τη θετική τους εμπειρία. Το 1992 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο κανονισμού για τα Ταμεία Ελασφάλισης. Δυστυχώς απεσύρθη το 2006 διότι δεν περπάτησε ούτως υπήν από νομοθετικής πλευράς. Και επίσης σε διάφορα κράτη-μέλη υπάρχει αυξημένος δυναμισμός αυτού του κλάδου, γιατί πάμε για το 25% της αγοράς ασφαλίσεων που έχουν και 70% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων του κλάδου. Άρα η ενιαία αγορά δεν μπορεί να αγνοεί το Ταμείο Ελασφάλισης. Πρόκειται για κάτι που πρέπει να τύχει προτεραιότητος. Έχουμε μόνο σε αυτούς τους βασικούς λόγους που μας δείχνουν ότι πρέπει να υπάρχει νομική ρύθμιση και τα ταμεία αυτά να μπορέσουν να σταθούν, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις στην εσωτερική αγορά, να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν, να αναπτύξουν τα στερεότυπα που έχουν στα κράτη-μέλη και να μπορούν να ανταγωνίζονται με όρους ε, ε, θεμητού ανταγωνισμού, μια που έχουμε τώρα αυτήν την ε, συγκυρία κρίση. Χρειάζεται να υπάρχει κάποια εφορία, χρειάζεται να υπάρχει κάλυψη για τους ε, ασφαλισμένους, γιατί όλο είναι και περισσότερο πρέπει να προσέξουμε πώς θα έχουμε κοινωνική οικονομία στις χώρες μας. Και επομένως ο ρόλος των ταμείων αυτών είναι σημαντικός για την ευρωπαϊκή οικονομία. Χρειάζεται επομένως να αποκτήσουν ένα ρυθμιστικό καθεστώς. Να, επομένως, γιατί γεννήθηκε αυτή η έκθεση από την Επιστροπή Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων. Είμαστε, επομένως, οι κυρίως αρμόδιοι. Βέβαια, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων διεξεδίκησε την, την αρμοδιότητα και θα αναλάβει η Νομική Επιτροπή τελικά την επί της ουσίας, ε, έκθεση. Όμως, Όσον αφορά την εργασιακή πτυχή των πραγμάτων και εμείς θα πρέπει να ασχοληθούμε με την πλευρά του θέματος που αφορά την απασχόληση. Τώρα νομίζω πρέπει να περάσει σκητάλη στους ε, ε, προσκεκλημένους μας. Έχουμε τον κύριο Ζεραντρέκ, τον πρόεδρο του ομίλου Μασίφ, κύριε Κάτριν Χόκ, ε, Γενική Γραμματεία του ΑΜΙΣ και τον κύριο Μπλεκ Ντασίλβα που είναι ο πρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως Άλλη Τα έχουμε τη χαρά πάντα να τους ακούσουμε. Να να Ελπίζω ότι όλοι επομένως θα κάνουμε κάτι για αυτή την κοινή ομαδική προσπάθεια. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Νομίζω ότι εσείς παρουσιάσετε την άποψή σας. Έχουμε και τρεις εμπειρογνώμονες και θα ήθελα εδώ να σας πω ότι ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και γι' αυτό ο καθένας θα έχει περιορισμένο χρόνο. Στη συνέχεια βέβαια θα, μπορείτε να, ε, ε, θα μπορούν οι παρουσιαστές να απαντήσουν και στις ερωτήσεις ε, των, των των επομένων ε, των Ευρωβουλευτών θα ρωτάνε. Ο, δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Ζεράρ Αντρέκ, πρόεδρο του ομίλου Μασίφ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ε, πρόσκλησή σας που δείχνει πόσο ενδιαφέρεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον τομέα της αλληλασφαλίσεως. Και η συγγήτρια άλλωστε αναφέρθηκε ε, και για να υπάρξει ένα καθεστώς ευρωπαϊκής αλληλασφάλισης από το 2005 έως το 2007 είχαν καταρτιστεί διάφορα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το 2010 υπήρξε μια γραπτή δήλωση. Το 2011 η έκθεση για τις ε, ε, αλληλασφαλίσεις και ε, γι' αυτό ε, θεωρούμε ότι στην έκθεση Μπανιέ αναφέρεται ε, η πράξη για την ενιαία αγορά. Αλλά ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς για να υπάρξουν όντως ισχύουσες αλληλασφαλίσεις στην Ευρώπη και να εξασφαλιστεί το μέλλον τους στην Ήπειρό μας. Διότι λόγω της κοινωνικοπολιτικής κατάστασης οποία επικρατεί. Γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να προωθηθούν στην Ευρώπη όλες οι επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας και βοηθούν την ανάπτυξη. Γι' αυτό και θα πρέπει ε, οι εταιρείε αυτές να συμβάλλουν εις τη δημιουργία κατά ε, ε, και εγκαθίδρυση των αξιών στην Ευρώπη στα πλαίσια των των στόχων της Ευρώπης του 2020 και να υπάρξουν τα αναγκαία μέσα για να μπορέσουν να αντιταχθούν ισότιμα στις κεφαλουχικές εταιρείες οι οποίες ήδη διαθέτουν ευρωπαϊκό καθεστώς. Γι' αυτό και σαν πρόεδρος της εταιρείας Massif που είναι αλληλασφάλισης θα σας παρουσιάσω τις αρχές της εταιρείας μας ε, και ε, σαν εκπρόσωπος των αλληλασφαλίσεων του ΖΕΜΑ, δηλαδή ε, των, της Γαλλίας, θα σας εξηγήσω πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη, τον κλάδο αυτό της ασφάλισης και να μπορέσουμε να τον ενισχύσουμε και να συγκροτήσουμε ευρωπαϊκά. Η Μασίφ καταρτίστηκε το 1960. Δεν έχει ούτε μετόχους, ούτε αμοιβέ ε, κεφαλαιουχικές, αλλά απλούστατα ε, προσπαθούμε να ρυθμίσουμε ε, τα ασφάλιστρα μέσω των κερδών και γι' αυτό θέλουμε να ενισχύσουμε τα ίδια κεφάλαια, να απομακρυνθεί ο οργανισμός από τις κερδοσκοπικές πρακτικές και να αποφευθεί η εκτροπή ε, και η μόχλευση. Εξού και ο ασφαλιζόμενος είναι και ασφαλιστής. Στην ε, ε, ε, κυβέρνηση μία ψήφος σημαίνει ένας εταίρος. Είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση και αποβλέπουμε στην κάλυψη των αναγκών των μελών και δημιουργία πλεονασμάτων τα οποία μπορούμε να επανα επενδύσουμε στο χώρο. Είναι δηλαδή οι στόχοι μας ταυτόσιμοι με αυτούς της Ευρώπης 2020 ε, και ε, η Γαλλία όπως ε, και η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ισπανία, η Ιταλία, οι κάτω χώρες και η Αγγλία και άλλες είναι από τους βασικούς πυρήνες τέτοιων αλληλασφαλίσεων και αποτελούν την βάση του θεσμού στην Ευρώπη διότι από 6-6,5 ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρώπη 3 3,5 χιλιάδες είναι αλληλασφαλίσεις χωρίς αυτό να εμποδίσει τον τομέα να καλυφθεί με έναν ενιαίο ορισμό και βάση των αρχών τις οποίες προανέφερα με συγχωρείτε που επιμένω για την δικιά μας οργάνωση, τη Μασίφ, η οποία είναι η πρώτη εταιρεία στη Γαλλία. Έχουμε πάνω από 5.000 ε, τέρους και μέλη ε, για τον τομέα της υγείας, της προλήψεως συλλογικής και ιδιωτικής, και προσφέρουμε ε, και τραπεζικές υπηρεσίες όπως και ασφάλειες ζωής. Ως εκ τούτου μπορούμε να καλύψουμε διάφορες λειτουργίες όπως αυτό γίνεται και σε άλλες χώρες όπως η Αγγλία όπου οι μεταφορές και οι υπηρεσίες υδροδοτήσεως καλύπτονται από τέτοιου είδους ε, ε, μορφές εταιριών. Σιγά σιγά λοιπόν η Μασίφ δημιούργησε ένα πολύ βασικό οργανισμό στην Γαλλία με πάνω από 5 εκατομμύρια μέλη, 9.000 ε, μισθωτούς που απασχολεί, έναν κύκλο εργασιών το 2011 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και επιπλέον καλύπτει ένα μεγάλο μέρος και των των ασφαλίσεων αυτοκινήτων ε, και των ασφαλίσεων κατοικίας ε, θα, στη συνέχεια ε, θα σας εξηγήσουμε γιατί πρέπει να αναγνωρίσουμε καλύτερα τις οργανώσεις αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν βασικούς παίκτες και παντού κατόπιν ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη κατόπιν του ανταγωνισμού και του κορεσμού των αγορών οι αλληλασφαλίσεις έχουν συγχωνευθεί και από 811 έχουμε 587 στην περίοδο 2007 σε 2010. Ε, για να αποφύγουμε λοιπόν την αποξένωση από αυτόν τον χαρακτήρα των αλληλασφαλίσεων που όπως συνέβη στην Αγγλία και στην Ισπανία, στη Γαλλία μπορούμε να δημιουργήσουμε μία μορφή η οποία εγγυάται τη διατήρησή τους και την ανάπτυξή τους. Εξού και ε, ε, δημιουργήθηκε μία εταιρεία των αλληλασφαλιστικών μήλων, η ΣΓΑΜ, η οποία ε, δεν έχει ίδιο κεφάλαιο και η Μασίφ μέσω αυτής μπόρεσε να συνεργαστεί και με τραπεζικούς οργανισμούς με μια πολύ μεγάλη συνεταιριστική τράπεζα την BCE ε, και ε, η ΣΓΑΜ ελπίζει ότι θα μπορέσει να συνεχίσει ε, από την ώρα που καταρτίστηκε το 2010 με δύο μεγάλους οργανισμούς την ΜΑΙΦ και την ΜΑΤΜΟΥΤ και ε, όλοι αυτοί ε, συγκεντρώνονται τώρα ε, γύρω από τις γκάμμα Μασίφ. Υπάρχουν διάφορα νομικά μέσα για τις οργανώσεις αυτών των ομίλων και αν θέλει κανείς να έχει διασυνοριακή ανάπτυξη μπορεί να χρησιμοποιήσει Α, τι, ε, τι, ε, ε μπορούν να προχωρήσουν αλλά όχι διασυνοριακά ε, διότι τότε θα υπάρξει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ε, όσες φορές προσπαθήσαμε διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις νομικώς Η Μασίφ λοιπόν έχει εγκατασταθεί στην Πολωνία, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία έχει καταρτήσει συνεργασίες ε, στα πλαίσια της Ρέζα με αντίστοιχη τύχες αλληλασφαλιστικές οργανώσεις γερμανικές στην 10 την στην Ιταλία με τη Unipol και στο Βέλγιο με την ε, ΠΕΒ ε και χρησιμοποιεί την ε, ελεύθερη παροχή υπηρεσιών κατά τρόπον ώστε ε, να προωθήσει ε, ένα νέο νομικό μέσα το οποίο ε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και εμποδίζει την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή προτείνουμε να υπάρξει μια αλληλασφάλιση ευρωπαϊκή η οποία να καλύπτει τις ανάγκες μας μας έχοντας αποδείξει ότι ο τρόπος επιχειρήσεώς μας πρέπει να στηριχθεί πιστεύουμε ότι στην Ευρώπη θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αντίστοιχους οργανισμούς όπως ε, η ΜΑΣΥΦ και να αναπτυχθούν πολύ γρήγορα διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομικός τρόπος να καταρτιστεί ένα τέτοιος όμιλος ευρωπαϊκός ή μία επιχείρηση ευρωπαϊκή και μόνο η ύπαρξη αυτού του βάθρου θα μπορούσε να επιτρέψει στις οργανώσεις να αναπτυχθούν στην Ευρώπη. Διότι για τις ευρωπαϊκές αλληλασφαλίσεις θα πρέπει να προωθηθούν παρεμφερείς δομές στις διάφορες χώρες για να διευκολυνθούν οι συγχωνεύσεις διασυνοριακά και να δημιουργηθεί ένα κοινό πλαίσιο που θα είναι ε, προσαρμοσμένο σε όλου και να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό σε ολόκληρο την Ευρώπη προς όφελος όλων των Ευρωπαίων ε, πολιτών. Ε, ε, ε, οι ορισμοί τους οποίους αντιμετωπίζουμε και πρέπει να έχουμε εφαρμόσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2014 μας υπενθυμίζουν ότι οι εταιρείε αυτές σήμερα είναι ε, εταιρείε ιδιωτικού δικαίου ανεξάρτητες και δεν επιδοτούνται. Μπορείτε να ολοκληρώνετε λέει η πρόεδρος παρακαλώ. Θα ήθελα να προσθέσω ένα στοιχείο σχετικά με τη στρέβλωση του ανταγωνισμού ότι με την νέα νομοθεσία ε, θα ε, καταστεί επιταγή να υπάρξει νομοθεσία σχετικά με την ε, Solvency 2 διότι προβλέπεται ρύθμιση εκεί η οποία καλύπτει τις ασφαλίσεις και αυτή τη στιγμή ε, μόνο δύο οργανισμοί είναι άμεσα ε, αναγνωρισμένοι στα πλαίσια της ε, ρυθμίσεως αυτής της φερεγγιότητος 2 και γι' αυτό θα πρέπει Αφενός να αναφερθούμε στην αύξηση των ιδίων πόρων, με συγχωρείτε. Ε, εσείς αντιλαμβάνεστε απλώς ότι οι συνάδελφοι ενοχλούνται εάν συνεχίζετε. Εγώ μπορώ να σας δώσω ακόμη 30 δευτερόλεπτα και όχι παραπάνω. Παρουσιάζω λοιπόν τα, ε, ε, τα συμπεράσματά μου. Νόμιζα ότι έχω 12 λεπτά, λέει ο μιλητής. Η Ευρώπη δεν πρέπει να εγκαταλείψει αυτόν τον βασικό τομέα που μπορεί να αποτελέσει πηγή αναπτύξεως και ε, απασχολήσεως είναι ε, οργανισμοί που δεν μπορούν ε, να μετακινηθούν γεωγραφικά και μία πηγή οικονομικής αξίας και καινοτομίας και μπορούν να αποδείξουν την ισχύ τους σαν ευρωπαϊκή αλληλασφαλιστική οργάνωση. Με συγχωρείτε αν ξεπέρασα την ώρα μου. Με συγχωρείτε που σας πίεσα, αλλά και εμένα αυτή είναι η δουλειά μου, λέει η πρόεδρος, και διότι δυστυχώς έχουμε ένα τόσο βαρύ πλαίσιο ε, και τόσο δύσκολη διαπραγμάτευση που σας προτείνω, εφόσον έχετε γραπτό στο κείμενό σας, να το δώσετε για να ε, τα βιβαστεί σε όλους τους συναδέλφους, οπότε όλοι θα έχουν το κείμενό σας και επιπλέον ε, έχετε ακόμη δύο λεπτά στη συνέχεια αν θέλετε να τονίσετε κάτι το οποίο είναι βασικό και θα θέλατε ε, να παρουσιάσετε. Τώρα θα δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή αλλά πριν από αυτό στον κύριο Γκρέγκορ Πόσνιακ ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας της ε, Association of Insurance Cooperatives in Europe. Πέστε μας λιγάκι τι είναι, διότι εγώ δεν πολύ κατάλαβα, λέει η Πρόεδρος, και θα έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Σας παρακαλώ μην τον υπερβείτε, διότι τότε ο κόσμος εκνευρίζεται και είναι δυσάρεστο. Εκτός μικροφώνου ο μιλητής. Uh, Ζητώ συγγνώμη, θα μιλήσω στα αγγλικά. Αγαπητή ε, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Συμφωνώ με την ευγνωμοσύνη του κύριου Άντρεκ για την πρόσκληση εδώ και αυτό αποτελεί απόδειξη της ε, διαρκούς υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μέλλον των ταμείων αλληλασφάλισης, όπως αναφέρεται σε εκθέσεις τα τελευταία δέκα χρόνια. Την περσινή καινοτόμο έκθεση για το ρόλο των ταμείων αλληλασφάλισης, τη σημερινή ακρόαση και το συνέδριο του Σεπτεμβρίου. Αποτελούν παραδείγματα όλα αυτά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζει τη σπουδαιότητα των τομέα των Ταμείων Αλληλασφάλισης. Η Ένωσή μας είναι ο οργανισμός εκπροσώπησης στην Ευρώπη όπως αναφέρεται στην ονομασία της ε, ε, συνεταιριστικών και ε, ταμιών ασφάλισης και ασφαλίσεων που ασφαλίζουν σήμερα σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις καθώς και παραδοσιακές δραστηριότητες ασφάλισης ε, σε μια εποχή όπου ο Δήμος Κορβανάς απομακρύνεται όλο και λιγότερο από τους τομείς αυτούς. Είναι όλο και πιο σημαντικό η παρούσα επιτροπή σε τέτοιες ε, εποχές ε, να αναφερθεί στο ζήτημα αυτό και να καλύψει το μέλλον και το πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. Δόθηκαν ήδη τα κυριότερα στοιχεία πάνω από 3 από τις 6.000 ασφάλειες στην Ευρώπη με μερίδιο αγοράς περίπου 25% στην Ευρωπαϊκή Ένωση 150, 160, 170 είναι δύσκολο να αποκτήσουν δικαιούχους ε, ε, στην Ευρώπη και πολλές χιλιάδες απασχολούμενοι. Το επιχειρηματικό μοντέλο των οικονομικών υπηρεσιών είναι ελκυστικό, ελκυστικό σε μακρονομικό πλαίσιο, διότι βασίζεται στην εγκύτητα στο μέλη μέσω δημοκρατικών διαδικασιών επικεντρωμένο στα μέλη και θέτει τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των μελών σε πρώτη προτεραιότητα όπως ανέφερα Πρόκειται για το τέλειο υποκατάστατο των όλο και λιγότερων κρατικών ενισχύσεων για βασικές ανάγκες των πολιτών. Επιπροσθέτως υπάρχουν μακροοικονομικά πλέον εκτίματα λόγω της παράλληλης ύπαρξης συνεταιριστικού και αλληλασφαλιστικού τύπου ε, ταμείων στην Ευρώπη διότι ο ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρηματικών μοντέλων αυξάνει, τι επιλογέ των πολιτών είναι ζωτικό για την αγορά, για την οικονομία και εν τέλει για τον Ευρωπαίο πολίτη. Τα ταμεία ελασφάλιση έχουν τι ιδιαιτερότητέ του ε, ορισμένε από αυτέ, αναφέρθηκαν ήδη, ε, ανήκουν στα μέλη του, ε, διαχειρίζονται από τα μέλη του, δεν υπάρχουν εξωτερικοί παροχή κεφαλαίου, συνεπώ δεν υπάρχουν μέτοχοι ανυπόμονοι που προσδοκούν αυξημένα κέρδη ε, στο επόμενο οικονομικό έτος. Ε, συνεπώς, λιγότερο βράχη πρόθεσμη οπτική των δραστηριοτήτων τους. Υπάρχουν συγκεκριμένοι δομή ισοζυγίων που χαρακτηρίζεται από την απουσία μετοχικού κεφαλαίου. Τα κέρδη αποτελούν τη μόνη πηγή κεφαλαίου μαζί με ε, εκκλήσεις προς τα μέλη στο πλαίσιο της αλληλεγγύης. Έχουν μια συγκεκριμένη δομή κόστους επειδή δεν βάζουν χρήματα στην άκρη για να πληρώσουν μερίσματα σε εξωτερικούς παραγωγούς κεφαλαίων. Λόγω της ε, εγκύτητάς τους με τους πολίτες, τα μέλη, τους ανθρώπους που ζουν, εργάζονται και δραστηριοποιούνται γύρω τους ε, έχουν συγκεκριμένες κοινωνικές ευθύνες. Φυσικά είναι νόμικες ε, δομές, το μοντέλο της αλληλασφάλισης και το νομικό πλαίσιο διαφέρει σε καθένα από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των 15, 16, 17 ουσιαστικά κρατών όπου υπάρχουν τα μία αλληλεασφάλιση. αλλά αρχίζουμε από τα κοινά χαρακτηριστικά από αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά προκύπτουν κάποιες προκλήσεις η χρηματοδότηση δεν θέλουν να μπουν στις κεφαλαίες αγορές ειδικότερα χρηματοδότηση της ανάπτυξης δεύτερον όρια όσον αφορά τις διασυνοριακές δραστηριότητες που μπορεί να είναι το αποτέλεσμα περιορισμών στις ευκαιρίες χρηματοδότησης, περιορισμών στις δυνατότητες συγχώνευσης σε εθνικό ή σε διασυνεροϊκό επίπεδο, στην ανάγκη σε ορισμένες δικαιοδοσίες δημιουργίας θηγατρικών αντί για ε, την ε, συνεργασία με ξένα μέλη και όπως είπα το μοντέλο δεν υπάρχει ή μάλιστα απαγορεύεται και σε ορισμένες χώρες ο σχηματισμός ομίλων είναι πολύ ε, πιο απίθανος για αυτές από ότι για τις ΕΠΕ μας μίλησε και ο κύριος Αντρέ για την εθνική δυνατότητα ομίλων ταμείων αλληλασφαλίσεων στη Γαλλία και αυτό αντικατοπτρίζεται από το γεγονός ότι το μοντέλο αλληλασφάλισης δεν υπάρχει σε πολλά κράτη-μέλη. Και έτσι τίθεται το ζήτημα της πανευρωπαϊκής αναγνώρισης. Η κυρία Μπάστο ίδια το ανέφερε στην εναρκτήρια ομιλία της. Ας δούμε τώρα ορισμένες από τις διαφορές στον τομέα της αλληλασφάλισης. Τα προβλήματα είναι τα ίδια, οι προκλήσει είναι οι κοινέ. Ωστόσο, αυτές οι προκλήσεις που αναφέρονται δεν αντιμετωπίζονται από όλα τα ταμεία αλληλασφάλισης ως προβλήματα παντού. Ορισμένοι τις δεν βλέπουν ως ευκαιρίες, ορισμένοι δεν ενδιαφέρονται και ορισμένοι δεν ενοχλούνται καθόλου από τους περιορισμούς. Άλλοι περισσότερο. Είτε διότι έχουν ελάχιστα διασυνοριακά συμφέροντα ούτως ή άλλως, διότι δραστηριοποιούνται τοπικά ή διακρίνουν λύσεις διαθέσιμες σε άλλους νομικούς τομείς. Εν μέρη, λόγω των διαφορετικών εθνικών μεθόδων, παραδόσεων, προσεγγίσεων όσον αφορά την αλληλασφάλιση, όλες αυτές οι διαφορές οδηγούν στη διαπίστωση ότι πολλές απαντήσεις, πολλές ανάγκες και πολλές διαφορετικές επιλογές υπάρχουν σε όλο το φάσμα του τομέα. Ως εκ τούτου οι λύσεις θα πρέπει να διαφέρουν. Αυτό το καθεστώς ταμείων αλληλασφάλισης που συντάχθηκε πρώτα απ' όλα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τους ενδιαφερόμενους αντιπροσωπευτικούς οργανισμούς είχαν αυτούς τις προκλήσεις στο νου τους. Σκοπός των σχεδίων κειμένου ήταν να αντιμετωπιστούν προκλήσεις που υπάρχουν από κοινού σε ολόκληρη την Ευρώπη στα ταμεία ελασφάλισης, στον ε, τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης, της ασφάλισης ζωής, σε άλλους τομείς επίσης. Ορισμένοι κάνουν μια έκκληση για ένα καθεστώ Ευρωπαϊκών Ταμείων Ελασφάλιση. Άλλοι επιθυμούν να λυθούν κάποια από τα ζητήματα που ανέφερα. Σίγουρα ο χρόνο εδώ δεν με επιτρέπει να μπω σε περισσότερε λεπτομέρειε για αυτέ τι προκλήσει. Τι ανέφερα ω επιμέρου σημεία. Και φυσικά είμαστε στη διάθεσή σα για να σα παρέχουμε περισσότερε πληροφορίε για αυτέ. Για να συνοψίσω, και δεν θα μπορούσα να είχα συνοψίσει καλύτερα από ότι του συντάκτε τη περσινή μελέτη που ανέθεσε η Επιτροπή Απασχόληση αυτού του Κοινοβουλίου. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στιβαρά επιχειρήματα ενίσχυση τη ασφάλιση. Υπάρχει μια έκκληση για διαφοροποίηση στον οικονομικό τομέα και όπω καταλαβαίνω αυτό συζητείται και στον τραπεζικό τομέα και σε αυτό το κοινοβούλιο και σε άλλους οργανισμούς ότι η ευρωπαϊκή τραπεζική δομή χρειάζεται διαφοροποίηση. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τον τομέα των ασφαλίσεων. Δεύτερον, υπάρχει μια μακροοικονομική επιμέρους πτυχή θα έλεγα για τις, τα ταμεία ελασφάλισης. Πολλοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν όλο και μεγαλύτερη ποιότητα ασφάλιση και κοινωνικές υπηρεσίες. Τρίτον, στο μέλλον βάσει των όσων μας λένε οι ερευνητές. Στο μέλλον οι ανάγκες θα μεγαλώσουν για όλο και περισσότερες εταιρείες με ε, βαθιά ριζωμένη κοινωνική ευθύνη στη δομή τους ώστε να παρέχουν φθηνή υψηλής ποιότητας, φθηνά υψηλής ποιότητας κοινωνικά συστήματα που θα συμμορφώνονται με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συντάκτες παρέχουν τρεις συστάσεις. Την πρώτη προς εμάς, προς τον τομέα της αλληλασφάλισης. Χρειαζόμαστε και συμφωνώ να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας και να διασπείρουμε την ιδέα της αλληλασφάλισης, της αξίας πυρήνα του οργανισμού μας. Δεύτερον, και αυτό το απευθύνω σε Ευρωπαίους και εθνικούς νομοθέτες και πολιτικούς να δημιουργήσουμε ε, συνθήκες ίσου ανταγωνισμού όπου οι παράγοντες στους οποίους βασίζεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των ταμείων θα έρθουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Και τελευταίο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η αλληλασφάλιση θα πρέπει να αναγνωριστεί περισσότερο. Και εδώ κάνω έκκληση εδώ στο Κοινοβούλιο, συμφωνώ με τη διαπίστωση ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο η αλληλασφάλιση θα πρέπει να αναγνωριστεί περισσότερο ως σημαντικός φορέας ε, άνισμα της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας. Εδώ κλείνω την ομιλία μου κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, Μπράβο σας που ε, το χρονικά όρια, τον περιορισμό. Ο επόμενο ομιλητή μα είναι ο Πέτρο Μπλεκδεσί, πρώτη IAIM, Διεθνού Ενώσεω Ελασφαλείας και θα του δώσω το λόγο, αλλά πρώτα-πρώτα. Θέλω να σα πω ότι δεν άκουσα την παρουσία σα, θα ακούσω όμω τι απαντήσει. Κύριε Πέτρο Μπλέκτα έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Περβόν Μπερές, πρόεδρε της Επιτροπής. Πριν προχωρήσω και σας παρουσιάσω τις θέσεις της Διεθνούς Ένωσης Άλληλα Ασφαλίζεως, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε, που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να σας ε, εξηγήσω εδώ τους λόγους για τους οποίους ε, προσπαθούμε να αναγνωριστεί στην Ευρώπη η ιδιοτυπία του κλάδου μας και να αποκτήσουμε κι εμείς ένα καθεστώς που να μας διέπει. Είναι επομένως μια τιμή να συμμετέχουμε στην προεδρική αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα σας τα πω όμως στα αγγλικά, γιατί είναι η γλώσσα ε, της ε, εργασίας μας εδώ και πολύ καιρό. Είναι επομένω οι ασφαλεί που είναι βαθιά ριζωμένε στην ευρωπαϊκή κουλτούρα, είναι πρόκειται ένα ολόκληρο σύστημα ασφάλιση και αν θεωρήσουμε ότι είναι το λίκνο του διεθνού πολιτισμού ε, Ευρώπη, τότε ήμασταν ε, ε, ω Ευρώπη τη Ασφαλίση, είναι υπόλοιπα προ μίμηση για όλο τον κόσμο, γιατί με την Ευρωπαϊκή Ένωση καλύψαμε όλε τι χώρε για δημοκρατία, για ελευθερία, όλου όσου σέβονται αυτέ τι αξίε και το κράτο ευημερία και πέραν των των διαφορών των κρατών μελών. Τελικά αυτή η πολυμορφία ήταν τελικά μια δύναμη και όχι αδυναμία και τελικά ε, όλα καταλήγουν και ξεκινούν βέβαια σαν δεσμεύσει ε, στον, στον άνθρωπο. Οπότε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να ανταποκριθούμε στι κοινωνικέ ανάγκε, να ξεπεράσουμε τι ε, ανισότητε και βέβαια το βασικό αρχή για όλα αυτά και το κλειδί είναι η ελληνική, η οποία είναι στην καρδιά του συστήματός μας, στην καρδιά του πολιτισμού μας οι αλληλασφαλίσεις, επομένως ε, είναι τέτοιες εταιρείε ε, προσω... Ε, αυτό μη κερδοσκοπικές, Όσον αφορά την επιλογή των κινδύνων, δεν έχουμε διακρίσεις και χρηματοδοτούμεθα με αλληλέγγυους τρόπους. Οι ασφαλίσεις βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης και της κοινωνίας των ασφαλιζόμενων ε, όσον αφορά τις απώλειες, ζημίες, ε, ε, τραυματισμούς και και όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, εμείς επομένως εκπροσωπούμε ως Διεθνής Ένωση Ασφάλισης πάνω από 160 δις Ευρωπαίους πολίτες που είναι ασφαλιστές τέτοιες εταιρείε, οι οποίες μπορούν να ασκούν τέτοιες ασφαλιστικές ε, δραστηριότητες ε, ε, όπου έχουν το βάρος να προστατεύουν τον εαυτό τους καταρχήν οι ασφαλισμένοι και επομένως να αναλαμβάνουν την ευθύνη, να καλύπτουν τις κοινωνικές τους ανάγκες, να καλύπτουν τους κινδύνους τους οποίους διατρέχουν με έναν τρόπο αηφόρο βιώσιμο και καλύτερο μπορεί να υπάρξει. Οπότε αυτό το οποίο εσείς έχετε πει για τον ε, ρόλο μας στον 21ο αιώνα είναι ότι τα ταμεία ελασφάλισης με αυτές τις αξίες δημοκρατίας διακυβέρνησης ε, ελασφάλισης και να μην χωρί να έχουν μετόχους είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά τα στήματα κοινωνικής προνοιάς και έχουμε αυτή τη μελέτη που δείχνει ότι για να μπορέσουμε να έχουμε αηφορία σε αυτά τα στήματα κοινωνικής προστασίας και φυραμιζόμενοι με του στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το οποίο χρειάζεται να λένε και περισσότερο οι, οι οικονομικά να ενεργούν με υπευθυνότητα, <clears throat> κάτι το οποίο να είναι βαθιά ριζωμένο σε αυτούς τους φορείς και οργανισμούς. Πέραν αυτόν η έκθεση σας λέει ότι το επιχειρηματικό μοντέλο αυτών των ανασφαλισμένων εταιριών είναι κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ, ιδίω τώρα με αυτή την συγκύρια τη κρίση, ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε τι αρνητικέ συνέπειε τη ε, κρίση προ του πολίτε και δεν φοβάμαι να σα πω ότι το επιχειρηματικό μα μοντέλο ε, είναι σταθεροποιητικό παράγον για τι οικονομίε μα και η σημερινή κρίση, επομένω, είναι μια μοναδική ευκαιρία για τα κράτη-μέλη αλλά και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να ενθαρρύνουν αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο σαν μια εναλλακτική και επομένως έτσι να έχουμε ε, καλύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Οπότε και αυτές οι εταιρείε ε, παίζουν ένα ρόλο πάρα πολύ σημαντικό ε, στα κοινωνικά. Όμως, το Ταμείο ασφάλισης επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγον και έχουν τη θέση τους στην στρατηγική για το 2020 της Ένωσης. Όμως εδώ τι χρειάζεται είναι να έχουμε μια ανάπτυξη αϊφόρο αλλά και ευφύ. Γιατί ξέρετε οι ταμείες ασφάλισης έχουν μέσα στα αγωνίδια τους την αλληλεγγύη. Ανέκαθεν αυτό. Ε, ήμασταν και θα ε, είμαστε παράγον οικονομικής ανάπτυξης. Και όπως είπαν οι προλαλήσαντες η ευρωπαϊκή οικοδόμηση θα πρέπει να καλύψει και εμάς γιατί δεν μας αναφέρουν όμως ε, οι συνθήκες, μας έχουν ξεχάσει. Όχι, γιατί έχουμε την ελευθερία υπαρχής υπηρεσιών, την ε, ελευθερία εγκατάστασης, που είναι πάρα πολύ βασικές και τελικά αυτές οι ελευθερίες θα πρέπει να ισχύσουν και για τα ταμεία ασφάλισης που θέλουν να αφήνουν σε άλλη ε, χώρα. Γιατί μας, μας ξέχασε ο νομοθέτης. Αυτό το οποίο σκέφτομαστε πάνω απ' όλα είναι ένα νομικό πλαίσιο, τόσο να μπορούμε να λειτουργήσουμε και να δουλέψουμε σε πνευματικό επίπεδο. Γιατί αν δεν υπάρχει τέτοιου είδου ε, νομοθεσία, πώ είναι δυνατόν να παρέσχουμε τι ε, υπηρεσίε μα. Μόνο με ένα τέτοιο νομοθέτημα, με ένα τέτοιο πλαίσιο θα μπορέσουμε να διδραματίσουμε τον ρόλο μα και έτσι να μπορέσουμε να είμαστε αναπόσπαστο τμήμα και να ωφεληθούμε από την ενιαία αγορά. Ιδάλλως, θα ε, είναι μια οπτασία, μια ψευδέστηση. Η αγορά και μια που τώρα έχουμε το, το γύρο του ποδοσφαίρου, τότε θα είχαμε δύο διαφορετικέ κατηγορίε στι ασφάλειες. Ορισμένοι θα παίζουν ε, στο Champions League που θα έχουν τι αθλητέ εγκατάσταση. και θα έχουν την ομοθεσία να τους διευκολύνει και επίση έχουν και τη δεύτερη κατηγορία εκείνοι επομένω οι οποίοι προσπαθούν και παλεύουν μόνοι του στην ε, αγορά. Επομένως, γι' αυτό και χρειαζόμαστε απελπιστικά το καθεστώς που θα μας διέπηκε, γιατί θα πρέπει να έχουμε δίκαιο ανταγωνισμό, το σούτο μάλλον, καθότι έχουμε τις, τους νομικούς από το Solvency 2. Θα πρέπει επομένω, αν θέλουμε να συμμορφωθούμε προς την οδηγία εκείνη, θα πρέπει να γίνουν ορισμένε αλλαγέ, ορισμένε ρυθμίσει, κυρίω όσον αφορά τα του ιδίου κεφαλαίου του, του εταιρικού. Εμεί προπήρχαμε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε τμήμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Επομένω, α έχουμε το θάρρο και το κουράγιο να στηρίξουμε αυτές τις ε, οντότητες να, τους, να τις πλαισιώσουμε όπως ε, αξίζουν και να τις βοηθήσουμε να ανθίσουν παντού στην Ευρώπη και έτσι αμφίβολα θα βοηθήσετε να ενδυναμωθεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. Και επομένως ε, η ευρωπαϊκή κουλτούρα, η ευρωπαϊκή κληρονομιά, η δάλος, λυπηρό να το διαπιστώνουμε, αλλά ένα τόσο σημαντικό τμήμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού τότε ε, είναι καταδικασμένο να φθήνει και τελικά να εξαφανιστεί. Και ας μην ξεχνούμε ότι η Ευρώπη ήταν και ακόμα είναι βασισμένη σε αυτό που είναι το ατού της, ο πλούτος της, τη διαφορετικότητα, την πολυμορφία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τους τρεις ε, προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες ε, στο πλαίσιο της έκθεσης ε, και της εργασίας της, της κυρίας Μπαστός. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά ωφέλιμα τα όσα ακούσαμε. Θα ξεκινήσω τη συζήτηση δίνοντας ε, πρώτα το λόγο στην κυρία Χαρκίνη και μετά τον κύριο Αρκάς. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και τους τρεις ομιλητές, όλους σας. Μιλήσατε πολύ ένθερμα και πολύ καθαρά και εκτιμούμε ιδιαίτερα την καθαρότητα αυτά. Έχω κάποιες ερωτήσεις και απλά Ήθελα να αναφερθώ στον τελευταίο ομιλητή όπου μιλήσατε για τον Ευρωπαϊκό Οίκο Δημοκρατία, Πραγματικά εύχομαι ορισμένοι συνάδελφοι που είναι απόντε αυτή τη στιγμή να ήταν εδώ και να άκουγαν τη δήλωσή σα αυτή. Μιλήσατε για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο. Αυτό προσπαθούμε να ασπαστούμε σε αυτή την Επιτροπή και χαιρόμαστε που βλέπουμε να το εκτιμά κάποιο διότι σε πολλού άλλου τομεί και σε πολλέ άλλε περιστάσει έχει απαξιωθεί. Έχω πέντε ερωτήσεις σχετίζονται με τους διάφορους ομιλητές. Πρώτα απ' όλα το ζήτημα της διαφοροποίησης που αναφέρθηκε. Θέλω να ρωτήσω, επειδή υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα σε νομίζω περίπου 17 κράτη-μέλη, μπορείτε να μας προτείνετε πού πρέπει να προσέξουμε, τι πρέπει να προσέξουμε στις προτάσεις μας, ώστε να μην έχουμε μη ανεπιθύμητα αποτελέσματα, διότι μια τέτοια διαφοροποίηση και μερικές φορές ίσως να νομίζουμε το μοντέλο ενός δύο κρατών μελών να ταιριάζουν σε όλα και πολλές φορές επικρίνεται έτσι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θα θέλαμε τη σκέψη σας γι' αυτό. Δεύτερον, ο συναδέλφος από την ΜΑΣΥΦ αναφερθήκατε σε συγχωνεύσεις και πώς προσπαθείτε να αποφύγετε την αποδυνάμωση της άλλης αναφέρατε το SGAM νομίζω που το πρόλαβε και που έχει εγκαθιδρυθεί. Θα μπορούσατε να μας το αναλύσετε λίγο. Είπατε ότι εντός ε, τριών ετών ε, μειώθηκαν τα ταμεία ασφάλισης κατά 300 θα συνεχίσει αυτό με τον ίδιο ρυθμό και ποιες προκλήσεις θέτει αυτό για τα ταμεία ασφάλισης όπως είπε ο συναδελφός σας ότι η εγκύτητα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του τομέα σας η τρίτη ερώτηση για τον δεύτερο ομιλητή ο οποίος μίλησε για κάλυψη αναγκών που δεν καλύπτονται αλλού μίλησε για την οπισθοχώρηση των κρατικών κονδυλίων συμβαίνει κάτι τέτοιο και για τα ιδιωτικά κονδύλια και θέτει αυτό ζητήματα για τα επιχειρηματικά μοντέλα σας και την κερδοφορία σας. Βλέπω ότι νεύετε με το κεφάλι, οπότε γνωρίζετε τι ρωτάω. Η τέταρτη μου ερώτηση αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο ταμείων αλλασφάλισης που εγώ γνωρίζω στη δική μου χώρα, την Ιρλανδία, το κίνημα Credit Union πιστοτικών ενώσεων. Υπάρχει σώρα κράτη-μέλη, αλλά σε πολλά καθόλου. Ένα από τα ζητήματα που έχει προκύψει οφείλεται στην οικονομική κρίση και στην απερίσκεπτη συμπεριφορά πολλών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως αποτέλεσμα το εκκρεμές έχει περάσει από τη μία πλευρά στην άλλη και με συνέπειες ε, για το κίνημα αυτό της πιστοτικής ένωσης ότι ορισμένοι οργανισμοί υφίστανται σημαντικές επιπτώσεις. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι οι νέες νομοθεσίες, οι νέες προτινόμενες νομοθεσίες και εθνικές που απορρέουν από την οικονομική κρίση. Γνωρίζετε κάποιες τέτοιες ε, για την οποία εσείς δεν ευθύνεσταν ή δεν γνωρίζατε. Η τελευταία μου ερώτηση, το Φερέγγιο τα δύο αναφέρθηκε αρκετές φορές. Ήθελα να ρωτήσω ζητήματα, προβλήματα που έχετε σε σχέση με τρέχουσα ή προτινόμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ξέρω ότι το τα 2 δεν σχετίζεται άμεσα με αυτήν εδώ την Επιτροπή, ωστόσο θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαρκάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας μιλήσω από πλευράς της πολιτικής μας ομάδας και να σας πω και η κυρία Ζίμπελη, η συγκίτρια, θα ήθελα να θέσει. Πολύ οικείο, πολύ αγαπητό, πολύ αγαπημένο θέμα είναι αυτό. Γιατί ξέρετε, έχω δουλέψει ως δικηγόρος σε μια τέτοια εταιρεία αλληλασφάλισης. Και έμαθα πολλά πράγματα. Και όπως είπαν οι συνομιλητές μας, έμαθα το πώς αυτό το πνεύμα της αλληλασφάλισης κατανέμει τον κίνδυνο στους περισσότερους ασφαλισμένους. Αυτό το είδος τους κινδύνους που διατρέχει ο καθένας από εμά. Και έτσι πολλαπλασιάζονται οι πιθανότητες, παρά το ότι ο καθένας μας είναι αδύναμος, να, να γινόμαστε πιο δυνατοί, μια που εν τη ενώση η δύναμη. Και αυτά τα διαπίστωσα και εδώ στον πολιτικό μου βίο. Δεν είναι μήπω και η Ευρώπη ένα τρόπο αλληλασφάλιση, που έχουν περισσότερε ευκαιρίε και λιγότερου κινδύνου. Και όταν και όταν χάνεται αυτό στην Ευρώπη, τότε βλέπουμε πόσο, πόσο, πόσο, πόσο άσχημα γίνονται τα πράγματα όταν χάνεται το πνεύμα της ε, ε, ελληνικής. Είμαστε κοινωνικά όντα. Ποτέ μόνοι μας χωρίς να συνεργαστούμε με άλλους δεν θα πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Τώρα, Ξέρετε, αυτή η νομική μορφή, αυτή η εταιρεία είναι πολύ αγαπητή σε σοσιαλιστές λόγω των ρεντισκών που έχει και γι' αυτό και θεωρούμε ότι θα πρέπει όντως να υπάρχει αντίστοιχα φιλική νομοθεσία της Ευρώπης. Για να δούμε τώρα κάτι που θα μας αφορά στο μέλλον για τη δουλειά μας. Πρώτα πρώτα, στα πλαίσια μιας τέτοιας φιλοσοφίας ε, κεφαλουχικών εταιριών. Βάση κεφαλουχική δεν είναι το πιο βασικό. Το πιο βασικό είναι η συμμετοχή. Ποιε είναι οι βασικέ απειλέ που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, ούτω ώστε μέσω του καθεστώτο να καλύψουμε τους κινδύνους από πλευρά διαχείρισης, ε, από πλευρά λογιστική, όλα αυτά τα οποία συντρέχουν και απειλούν τους σκοπούς της εταιρείας θα ήθελα επομένω να μάθω εσείς οι τρεις προσκεκλημένοι μας τι περιμένετε από μας εδώ στο Κοινοβούλιο. Πώς θα γίνει να προωθήσουμε αυτό το οποίο εκπροσωπείται και είναι τόσο θεμελιώδης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ε, Πρόεδρος, πριν λάβει το λόγο κύριε Μπάστος, θέλει άλλο το λόγο. Όχι. Εγώ ίδια θα λάβω όμως το λόγο. Και θέλω να τους πω το εξή στους προσκεκλημένους μας. Μπορεί ο καθένας από εσά να μας πει τρεις λόγους για τους οποίους θα πρέπει να αποκτήσουμε ένα τέτοιο καθεστώς για το Ταμείο Δεύτερο ερώτημα. Ποιες είναι οι τρεις προτεραιότητες που θα πρέπει να καλύψει αυτό το καθεστώς ή τα τρία βασικά εμπόδια για τη συγκρότηση μιας τέτοιας εταιρείας που πρέπει να καλύψει επίσης το καθεστώς. Είπα ότι θα πρέπει εκτός καθεστώτος να βιληθούν τα πράγματα. και οι, και οι ασφαλιστικές εταιρείες να μπορούν να παράσχουν τις υπηρεσίες τους. Τι θα πρέπει ο μέρος να γίνει. Δεν ξέρω ποιος θα απαντήσει, αλλά εάν αφού μιλούμε για ευρωπαϊκό καθεστώς. Όταν κάνει, ξέρετε, η Επιτροπή ένα σχέδιο οδηγίας ή κανονισμού, προσπαθεί να διαπιστώσει τις επιπτώσεις του νομοθετήματος. Τα ξέρετε τώρα τα επιχειρήματα που υπάρχουν υπέρ των ελασφαλίσεων, αλλά ένα επιχείρημα γιατί πρέπει να αποκτήσουμε καθεστώς είναι που νομίζω ο κύριος Ντασίλβα το ανέφερε όταν θέλουν αυτές οι ελασφαλίσεις να παρεύουν κάπου εκτός χώρας προέλευσης αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Θα πρέπει να απαντηθεί αυτή η ερώτηση, αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Αυτά ήθελα να σας ρωτήσω. Αλλά φαντάζομαι ότι και η κυρία Μπάστος έχει να θέσει σημαντικά ερωτήματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες αλλά όλους ε, που συμμετείχαν και ε, έχουν διατυπώσει και τροπολογίες και για τις ενδεχόμενες μελλοντικές τροπολογίες. Καταρχήν, σχετικά με τις παρουσιάσεις, η ε, βασική ιδέα είναι ότι η αλληλασφαλίσεις ε, βασίζονται στην αλληλεγγύη και είναι η βάση του ευρωπαϊκού σοσιαλιστικού και κοινωνικού προτύπου ε, για τη χρηματοδότηση και την ασφάλιση και έτσι μπορούν να εναρμονίσουν την νομοθεσία στα κράτη-μέλη για να βρεθεί ο ελάχιστος κοινό παρανομαστής για τα δικαιώματα όλων. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε τι πρέπει να μας απασχολήσει και πώς μπορούμε εμείς να επέμβουμε. Αυτό ρώτησαν και οι συνάδελφοι ε, τους εμπειρογνώμονες. Ποιο είναι το βασικό στοιχείο στο οποίο πρέπει να εστιαστούν οι Ευρωπαίοι. Ποιος είναι ο ελάχιστος κοινό παρανομαστής ε, το, που πρέπει να απασχολήσει τον Ευρωπαίο νομοθέτη κατά τρόπον ώστε να μην κινδυνεύσει το ισχύον ε, ασφαλιστικό πρότυπο και υπό αυτές τις προποθέσεις ποιο θα είναι το προσόν του να υπάρχει ο κοινός ο παρανομαστής για να λειτουργήσουν αυτές οι ε, ε, ασφαλιστικές ε, οργανώσεις. Υπάρχει και το θέμα της ε, επικουρικότητος που πρέπει να μας απασχολήσει, ιδίω όσον αφορά την εμπλοκή του δημοσίου τομέα, των μεταφορών, της υγείας κτλ. Ένα άλλο θέμα το οποίο νομίζω ότι τίθεται σαν αρνητικό για τη δημιουργία Ενό ενός ευρωπαϊκού ενιαίου καθεστώτος είναι ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και γι' αυτό ορισμένοι αντετάχθησαν στην ύπαρξη αυτού του καθεστώτος και του κανονισμού. Ε, θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε εσείς σαν εμπειρογνώμονες που, ε, που υπάρχει έλλειψη νομοθεσίας η οποία μπορεί να εμποδίσει την πρόθεση σχετικής νομοθεσίας στην Ευρώπη. Ακολουθούμε την ίδια σειρά, εάν θέλετε. Ο κύριος ε, Ζεραλάντεκ. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω σε μερικές από τις ερωτήσεις, διότι στο σύνολο δεν θα τα καταφέρω. Το ζήτημα της διαφοροποίησης ε, αποτελεί ένα εμπόδιο για μια ευρωπαϊκή, ένα ευρωπαϊκό ταμείο ασφάλισης. Οι εργασίε που έχουμε κάνει δείχνουν ουσιαστικά το αντίθετο. Πρόκειται για πλούτο. Αναγνωρίζονται, έχουν τις ίδιες αρχές, τους ίδιους προσανατολισμούς ε, τα ταμεία ασφάλισης. Τώρα για την πρώτη ερώτηση, ποιοι είναι οι φραγμοί, τα εμπόδια σε ορισμένες χώρες. Είναι μια πολύ παλιά παράδοση σε άλλες ε, χώρες όπως είπε η κυρία η δεν υπάρχει τίποτα η πρώτη συνθήκη λοιπόν είναι να μην έχουμε ένα περιοριστικό πλαίσιο αλλά να αναφερθούμε σε μια σειρά αξιών κατά την απόψή μου οι αξίες είναι πολύ απλές ισότητα μεταχείρισης, διακυβέρνηση, εγκύτητα η διακυβέρνηση λοιπόν θα πρέπει να ανήκει στα μέλη. Αυτό είναι το πλεονέκτημα, να διατηρήσουμε αυτό το πνεύμα διακυβέρνηση. Επίσης η συμμεταχείριση και η εγκύτητα και η κάλυψη πρέπει να πούμε κοινωνικών αναγκών. Συχνά ξεχνάμε, τώρα απαντάω λίγο μαζικά σε όλες τις ερωτήσεις, ε, θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι αυτή τη στιγμή τα Ταμεία Αλληλασφάλισης καλύπτουν ε, τα κενά των κρατών ε, σε ορισμένους τομείς, ιδίως της υγείας και στον κοινωνικό τομέα για τον ίδιο λόγο και την αποδέσμευση του ιδιωτικού τομέα που δεν ε, έχει κερδοφορία σε αυτόν τον τομέα και αποσύρεται. Έχουμε λοιπόν ένα ρόλο και ζητώ συγγνώμη τώρα που υπερβάλλω κλείνουμε τρύπες ουσιαστικά και γι' αυτό είναι σημαντική η παρουσία μας σε αυτόν τον τομέα. Μιλώντα λοιπόν για ένα πλαίσιο, πρέπει να έχουμε υπόψη μα τις τοπικές συνθήκες και πραγματικότητες και να επιθυμίζουμε τις κοινέ μας αρχές. Ε, θα μπορούσαμε να τι χρησιμοποιήσουμε αυτές ως ε, λογοτυπό μα ουσιαστικά. Ε, το, το σχέδιο βασίστηκε σε χαρακτηριστικά κοινά λειτουργία στην Ευρώπη όπως ε, εντοπίστηκαν λαμβάνοντας ε, υπόψη τις ιδιαιτερότητες αναχώρα. Αυτό έχει επικυρωθεί, έχει συμπεριληφθεί στην έκθεση και δεν ε, υπάρχει αντίθεση από κανένα μέρος για αυτό το θέμα. Όσον αφορά την ΣΓΑΜ, δεν μιλάμε για εργαλείο συγχώνευσης, είναι το αντίθετο, είναι εργαλείο προσέγγισης των ταμείων αλληλασφάλισης που θέτουν ε, σε κοινή χρήση μια σειρά έργων. Αντίθετα από άλλα εργαλεία όπως το GIE που επιτρέπουν την, τον κοινοχειρισμό ορισμένων δραστηριοτήτων, η ΣΓΑΜ επιτρέπει ε, κοινή χρήση για πόρων για νέα έργα, αλλά δεν αποτελεί συγχώνευση. Είναι το αντίθετο Δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη συγχώνευση. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εάν το επιθυμείτε μπορούμε να σας δώσουμε και προς τις πληροφορίες επί του θέματος. Όσον αφορά τη μείωση των ταμείων αλληλασφάλισης έχουμε διαπιστώσει όντω τη μείωση του αριθμού ο οποίος δεν σημαίνει απαραίτητα μείωση των μελών, του αριθμού των μελών. Συχνά πρόκειται για μια μείωση που σχετίζεται με φαινόμενα ε, συγκέντρωσης ε, ταμείων. Ε, αυτό φαίνεται στην Ευρώπη. Η Φερεγγιώτα αποτελεί απειλή γι' αυτό. Έχει ως αποτέλεσμα ότι ορισμένες απαιτήσει δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν από τα, ορισμένα ταμεία ελασφάλισης λόγω μεγέθους τους. Η μείωση των ταμείων, για παράδειγμα, στην Αγγλία αποτέλεσε δηλαδή το τέλος αυτών των ταμείων υπάρχει ένας κίνδυνος ε, διότι είπα ότι διαφυλάσσουμε την απασχόληση στη Γαλλία ο τομέα τη κοινωνική πολιτική, δηλαδή των ταμείων αλλασφάλιση, δημιουργεί τα τελευταία χρόνια διπλάσιε θέσει απασχόληση από ό,τι δημιουργούνται αλλού. Από τον υπόλοιπο παραδοσιακό, ε, θα έλεγα, καπιταλιστικό τομέα. Η μείωση λοιπόν αυτών των ταμείων ε, αλλασφάλιση ε, εξαφάνισε πολλές θέσεις εργασίας. Ε, θα σταματήσω εδώ και θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους μου, αλλά αντιλαμβανόμαστε ακόμη και σε χώρες ε, ισχυρής μείωσης τα ασφάλισης, το αντιλαμβανόμαστε. Αυτοί που υποφελούνται τελικά, δηλαδή οι κοινωνίες, οι καταναλωτές, είδαν τα ασφαλιστικά τους θέλουν να αυξάνονται και την επανικοδόμηση τέτοιων μορφών. Αναφέρεται την Ιρλανδία, αλλά σήμερα έχουμε ένα φαινόμενο εξισορρόπησης προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Προσνιάκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλές είναι ερωτήσεις πρέπει να απαντήσω και θα επιταχύνω. Ξέρετε, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της πολυμορφίας είναι η ιστορία, η νομική οι παραδόσεις, το πώς γίνεται αντιληπτή η υπαρξία λειτουργία των ταμείων ασφάλισης. Το τερικό δίκαιο δηλαδή το οποίο διέπει κάποιες, ε, κάποιες ε, κάποιες, κάποιες εταιρείε και εδώ το δίκαιο το οποίο διέπει τα, τα ταμεία ασφάλισης είναι δίκαιο πάρα πολύ συγγενές στο εταιρικό δίκαιο. Ε, στην Ιταλία, Φερρυπίν, ε, είναι εταιρείε αστικού δικαίου με δικό του καταστατικό. Σαν να αυτών των ιστορικών λεπτομεριών ε, υπάρχει διαφορετική αντίληψη εκεί για το τι είναι το Ταμείο Ελλασφάλισης. Επομένως, η ελεγγύη υπάρχει, όμως το θέμα είναι, είναι το θέμα της ανεξαρτησίας, το κοινωνικό πρότυπο, ο μη κερδοσκοπικό βασικά χαρακτήρα τους, ενώ όλα αυτά. Και έτσι κάποιες ε, εθνικέ κοινότητε φοβούνται ότι θα χάσουν με την εναρμόνιση τα εθνικά τους χαρακτηριστικά. Και ξέρω πολύ καλά ότι ο φόβος είναι, όποτε συζητεί τέτοια πράγματα η Ευρώπη, ότι θα επηρεαστούν οι εξελίξεις και όλες οι χώρες τώρα θεσπίζουν νέο ασφαλιστικό δίκαιο. Οπότε και οι αντίστοιχοι υπουργοί θα ήθελαν να αλλάξουν το καθεστώ που διέπει το Ταμείο Ασφάλεια στη χώρα του, ε, το θετικότερα ή προς αρνητικότερα, γιατί ε, έχουν χτυπηθεί από αυτόν τον ε, σκεπτικισμό, την, την υποψία σε σχέση με αυτές τις εταιρείες και αυτά τα οποία τώρα παρέχουν. Τώρα όσον αφορά τη φερεγγιότητα 2, το Solvency 2, το πρόβλημα είναι όχι η νομική μορφή, αλλά το μέγεθος. Και μιλώ για μικρομεσαίες, ελασφαλιστικές ή ε, αυτό αφορά και τις μικρομεσαίες ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι όλο θέμα αναλογικότητας καθαρά. και το θέμα των ομίλων ασφαλιστικών ε, τέτοιων εταιριών δεν επιλύεται από το Solvency 2. Κύριε Σέργα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σα λόγια, ε, για το πόσο είστε προσιλωμένος σε αυτές τις αξίες που τα διακυβεύονται και αυτό είναι αλήθεια το οποίο αφορά και τις ασφαλιστικές και τις ε, ασφαλίσεις κοινωνικής προνοίας για, για, για όλους τις ασφαλίσεις τέτοιου είδους παντού, παντού. Νομίζω ότι όλοι μας τονίσαμε πόσο σημαντικές είναι αυτές οι αξίες. Και σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Κύριε Πρόεδρε, Μπερές. Από τι αντιλαμβάνομαι. Βασίλειο για να υπάρξει ένα τέτοιο καθεστώς είναι το θέμα της αναγνώρισης. Το Ευρωπαϊκό Σήμα του ΣΥΠΗΝ και εδώ επανέλθω στη, στα όσα είπε η κυρία Μπάστος. Η διευκόλυνση του να αναπτύσσουν δραστηριότητε διασυνοριακά. Είναι πρόβλημα επομένω ο φόβος του ρυθμιστικού πλαισίου από κάποιο τέρας των Βρυξελών, α πούμε. Πάντως λέει ότι δεν χρειάζεται εναρμόνιση. Δεν χρειάζονται τις βασικές ελευθερίες της κοινή αγοράς. Το οποίο φυσικά μας παραπέμπει στα σωπή κυρία Μπάστος για τις διασυνορικές υπηρεσίες παρέχονται και σε όσο είπατε εσείς κύριε Μπέτας σε ευρωπαϊκό επίπεδο κινούμεθα για αυτές τις προκλήσεις ε, στις δυνατότητες που προσφέρονται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και το θέμα είναι κατά πόσον θα πρέπει, μπορεί η Ευρώπη να αντιμετωπίσει με το καθεστώς αυτά τα προβλήματα. Τα θέματα είναι γνωστά, έχουν επισημανθεί, είναι κοινά. Το θέμα είναι βέβαια ποια είναι η πιο σωστή προσέγγιση Και ακριβώ γι' αυτό και το συζητούμε τώρα όσον αφορά την κοινή αγορά. Ναι. Είναι αλήθεια ότι αν υπάρχουν δυσνορικές ρυθμίσει, αυτό θα ωφελήσει τι ασφαλιστικέ συμβάσει. Δίνονται ευκαιρίε, πολλέ από αυτέ μπορούν οι ασφαλίσει να εκμεταλλευτούν. Όσο αφορά κάποια πρότυπα που δεν είναι γνωστά σε κάτι μέλη. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε αντιρρήσεις στο να συγκροτηθούν τέτοιες εταιρείε. Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει αδιαφορία. Περισσότερο έχουμε σκεπτικισμό, έχουμε δισταγμό εκεί που ήδη υπάρχει ένα ριζωμένο, δοκιμασμένο μοντέλο. σε ένα μοντέλο το οποίο θεωρείται ότι δεν βοηθάται από όσα έχουν ρυθμιστεί πώς θα ρυθμιστούν τώρα σε σχέση με αυτά που ρύθμισε πριν 20 χρόνια η Κομισιόν πριν 5 χρόνια ο, ο κλάδος. Τώρα όσον αφορά το, το, το, το Solvency 2 βλέπουμε να υπάρχει εδώ πέρα κάποιο είδους προστατευτισμό ούτως ώστε το να ανοιχτεί αυτή, αυτή η ρύθμιση εκεί που απλώς έχουμε συνεταιρισμούς ε, τι θα γίνει. Επομένως, αυτό έχει να κάνει και μας όπως είπε η κυρία Μπάστος που φοβάται ότι εάν οι αντιλασφαλίσεις μπουν εκεί που δεν υπάρχουν τέτοιες εταιρείες ακόμα, το τι θα γίνει. Τότε είναι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα από, την ύπαρξη των εταιρείων σε αυτές τις αγορές για πρώτη φορά και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Comecei em Προσπαθήσω να ολοκληρώσω στα πορτογαλικά που είναι η μητρική μου γλώσσα. Εγώ πιστεύω ότι οι ερωτήσεις που τέθηκαν, παρότι ορισμένες φορές φαίνονται ασύνδετες, συνδέονται μεταξύ τους ουσιαστικά και με το ουσιώδες ερώτημα τα ταμεία αλληλασφάλισης από το κομμάτι του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Η Ευρώπη αποτελείται από πολλές χώρες και στη συνέχεια όλο διευρύνεται και σήμερα είμαστε πλέον 27 χώρες. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα έχουμε ένα κοινωνικό μοντέλο το οποίο δεν είναι απολύτως εφαρμόσιο ή επεκτάσιμο που δεν υπάρχει σε όλες, όλες τις χώρες αλλά μόνο σε ορισμένες. Αν εμείς επιθυμούμε μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, πρέπει πραγματικά να στοχεύσουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική αλληλεγγύης και το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο βασίζεται στην αλληλεγγύη. Συνεπώς, εάν εμείς ε, το μοντέλο αυτό αλληλεγγύη κοινωνική προστασίας το φέρουμε στις χώρες που δεν το γνωρίζουν, δεν γνωρίζουν αυτή τη μορφή αλληλεγγύης. Ενισχύουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αυτό το ερώτημα οδηγεί σε μια άλλη πιο τεχνική πτυχή. Γιατί τα ταμεία ασφάλιση και αναφέρομαι κυρίως τα ταμεία ασφάλιση για την υγεία που αυτά τα ταμεία ασφάλιση που κατά βάση έχουν εθνικές ρίζες θα έπρεπε να μετακινηθούν σε άλλες, να μεταφερθούν σε άλλες χώρες που δεν γνωρίζουν αυτό το μοντέλο ή που το χρησιμοποιούν με μια πιο αδύναμη μορφή. Τα ταμεία ασφάλιση, σε παραλαμβάνω, βασίζονται στην αλληλεγγύη και εμεί θέλουμε να ε, παρέχουμε προστασία των πολιτών και σε άλλε χώρε, Αλλά αυτά τα ταμεία ασφάλισης ε, απευθύνονται σε αγορές με ε, νομικούς κανονισμούς, ε, απαιτήσεις, κυρίως όσον αφορά την απαιτήση για ίδια κεφάλαια, για να μπορούν λοιπόν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε αυτή την πιο διευρυμένη αγορά. Ταυτόχρονα με άλλους τύπους οργανισμών που έχουν κεφαλαιακούς κανόνες και δυνατότητες πρόσβασης στις κεφαλαίες διαφορετικές, τα Ταμεία Ασφάλισης στην παρούσα στιγμή Θέλοντας να δραστηριοποιηθούν σε άλλες χώρες, χρειάζεται να έχουν ένα καθεστώς ευρωπαϊκό Ταμείο Ασφάλισης που θα τους επιτρέπει την μετακίνησή τους όχι μόνο εντός της χώρας τους αλλά και σε άλλες χώρες αξιοποιώντας τις ε, οικονομίες κλίμακας, ενισχύοντας έτσι τα κεφάλαια τους δύο, την ενισχύοντας τα ίδια τους κεφάλαια, τις δικές τους δομές και τη δική τους αηφορία και βιωσιμότητα έτσι ενισχύεται προφανώς και η ελληνική μεταξύ των διαφορών χωρών. Εδώ ωστόσο τέθηκε ένα ερώτημα από την αξιότιμη κυρία Ρετζίνα Μπάστος είτε τα ταμεία αλληλασφάλισης που ήδη υπάρχουν σε ορισμένες χώρες για ποιο λόγο χρειάζονται καθεστώς δικό τους. Αυτή η ερώτηση τέθηκε από πολλά μέλη. Τα ταμεία ασφάλισης, ναι, λειτουργούν σε ορισμένες ε, χώρες αλλά υπό διαφορετικά νομικά καθεστώτα. Ο κίνδυνος λοιπόν που τίθεται όσον αφορά τα ταμεία ασφάλισης και έχει αναγνωριστεί αυτός ο κίνδυνος ε, στη μελέτη που έχει επιτευχθεί μετά από εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κίνδυνος αυτός είναι ότι τα ταμεία ασφάλιση μπορεί να χάσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους όταν ε, μεταβούν σε άλλε χώρες για να διευρύνουν τι δραστηριότητε του όταν σε αυτές τις χώρες υπάρχουν διαφορετικές νομικές μορφές για τις ε, κερδοφόρες εταιρείες. Εκεί τα ταμεία ασφάλιση χάνουν τα χαρακτηριστικά τους. Και έτσι με κάποιο τρόπο ουσιαστικά χάνουν το χαρακτήρα της αλληλασφάλισης. Και αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Εμείς θέλουμε να το καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε ακριβώς αυτό έχοντας ένα ευρωπαϊκό καθεστώς Ταμείο ασφάλισης θέλουμε να αναγνωριστεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο διότι εσπιζόμενοι αυτό εμείς διεκδικούμε τη δική μας ε, ε, παρεμβολή ως μέλη για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς διότι διαφορετικά θα απολέσουμε τα χαρακτηριστικά μας αν πράξουμε διαφορετικά για μας είναι θέμα ζωής ή θανάτου το καθεστώς των ταμείων αλλασφάλισης θα πρέπει να είναι ένα διαβατήριο που θα μα επιτρέπει να πάμε σε άλλες χώρες. Έχοντας έτσι λοιπόν ένα σύνολο κοινών χαρακτηριστικών, πολλά μεν εθνικά μοντέλα, αλλά σίγουρα το καθεστώς ε, ε, το ευρωπαϊκό δεν θέλει να δημιουργήσει επικαλύψεις. Ένα τέτοιο καθεστώς θα είναι σίγουρα ένα προαιρετικό εργαλείο δεν θα επιβληθεί σε σχέση με τις εθνικές νομοθεσίες. Αποτελεί απλά ένα σημείο αναφοράς, μια δυνατότητα που παρέχεται στα ταμεία να μπορούν να κυκλοφορήσουν στον ευρωπαϊκό χώρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι σαφέστατα επιχειρήματα για να υπάρξει μια ευρωπαϊκή ρύθμιση. Υπάρχει άλλη μια ερώτηση που θα ήθελα να κάνω επιπλέον, ο, αν το θέμα που συζητάμε είναι επίκαιρο. ή εργαζόμαστε με διαφορετική φιλοσοφία. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει ε, ένα νέο πεδίο, απλούστατα ότι υπάρχει μία πολιτική κινητοποίηση για να προχωρήσουμε κατά τρόπον ώστε μετά την έκθεση της κυρίας Μπάστος μαζί με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων βάσει της μελέτης την οποία καταρτήσαμε πέρυσι να μπορέσει να προχωρήσει το θέμα αυτό το οποίο είναι πολύ ουσιαστικό τόσο για τα, στα πλαίσια της ρυθμίσεως φερεγγιότητα 2 όσο και στο ότι παραμένει ένα θέμα επίκαιρο που χρήζει ρύθμιση. κυρία Μπάστος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επαναλαμβάνω τα συγχαρητήριά μου και τις ευχαριστίες μου προς τους εμπειρογνώμονες και στους συναδέλφους που παρενέβησαν κατά την ακρόαση και ήθελα να πω ότι όλοι εμείς ουσιαστικά καταλήγουμε στα ίδια συμπεράσματα, δηλαδή την ανάγκη ευρωπαϊκής νομοθεσίας που να προβλέπει ένα ευρωπαϊκό καθεστώς για τα ταμεία αλληλασφάλισης όχι όμως μόνο για να διαφυλάξουμε το συγκεκριμένο πνεύμα αλληλεγγύης και δημοκρατίας και οργάνωσης των Ταμείων Αλληλασφάλισης αλλά και για να δώσουμε μια σημαντική όθηση στην εσωτερική μας αγορά ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτό το τομέα μια νέα εποχή σε μια στιγμή όπου η Ευρώπη χρειάζεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κοινωνική προστασία και την απουσία αποκλεισμών. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλουμε να μεταδώσουμε με κάποια προσοχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θέλουμε να πιέσουμε για επιτάχυνση ενός καθεστώτος. Θέλουμε να υπάρχει μια ελάχιστη εναρμόνιση ώστε οι εθνικές νομοθεσίες να μπορέσουν να υιοθετήσουν αυτό το καθεστώς χωρίς αρνητικές επιπτώσεις ε, ε, στις παραδοσιακές ε, μορφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναφέρουμε ε, το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή οι τροπολογίες μέχρι τις 11 ε, του Ιουλίου, 12 το μεσημέρι και εν ονόματι όλων μας θέλω να ευχαριστήσω τους τρεις προσκεκλημένους μας, να τους πούμε ότι η πόρτα μας είναι πάντοτε ανοιχτή, εάν πέραν τη σημερινή συζητήσεω έχουν συγκεκριμένες προτάσεις που θέλουν να μας διαβιβάσουν και ε, χάρη σε αυτή την έκθεση κατά πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορέσουν να προωθήσουμε ενδεχομένω και άλλα μελλοντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ερχόμαστε λοιπόν στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης τώρα το οποίο μας οδηγεί στο να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κοζά για να κοιτάξουμε τις τροπολογίες ε, σύμφωνα με ε, το ε, κανονισμό 444 στα πλαίσια του κοινού στρατηγικού πλαισίου για το Ταμείο Συνοχής.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 ξεκινήσω την παρουσίασή μου, θα σας δώσω μερικά στατιστικά στοιχεία. Έχουμε... Για να παρουσιάσω την έκθεσή μου πρέπει να πω ότι έχουμε πολλές τροπολογίες, άρα ευθύς εξ αρχής πρέπει να ισχύσουν διάφορες ε, συμβιβαστικές τροπολογίες. Εξού και σήμερα έστειλα ε, ε, μία πρόταση στο σκιώδη εισηγητή με συγχωρείτε, ε, γύρω μου γίνεται χάος και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Μπορώ παρακαλώ να παρακαλέσω όσους θέλουν να φύγουν να βγουν σιωπηλά και να κάνουν συζητήσεις στις εκτός αισθούσεις ε, και αν θέλουν στη συνέχεια να μπορέσουν να επανέλθουν. Τώρα κύριε εισηγητά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επανέρχομαι λοιπόν, εάν δεν έχετε αντίρρηση και θα σας πω ότι έχουμε ε, πάρα πολλές τροπολογίες όπως ανέφερε η Πρόεδρος και προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές προτάσεις τις οποίες στείλαμε. Πρόκειται για 55 συμβιβαστικές τροπολογίες ε, που έχουν αποσταλεί στους κοιόδης εισηγητές και πρέπει να σας πω ότι μέσω αυτών των συμβιβαστικών τροπολογιών ε, καλύπτουμε περισσότερες ε, ε, προ τροπολογίες που έχουν υποβάλει 15 ευρωβουλευτές και αντιλαμβάνεστε ότι κοινωνικά η Επιτροπή μας εμπλέκεται πλήρως και αποβλέπει στη βελτίωση των συνθήκων ζωής των μισθωτών εκτού, εξού και καταλήξαμε σε 55 συμβιβαστικές τροπολογίες προς το παρόν όμως είναι, ε, είναι απλώς προτάσεις για συμβιβαστικές τροπολογίες διότι μέχρι στιγμής δεν έχω συναντηθεί με τους χιώδεις εισηγητές και ε, δεν νομίζω Νομίζω πάντως ότι θα υπάρξει πόλωση στην προσέγγιση μας και πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε πολύ στενά για τη συνέχεια. Έχουμε όμως δυσκολίες για το δεύτερο τμήμα, διότι πλέον αυτού έχουμε πάρα πολλές προτάσεις, δηλαδή είμαστε συνομοθέτες ε, μαζί με την ε, Επιτροπή Περιφερειών και υπάρχουν τέσσερις ε, πολιτικές ομάδες που έχουν διατυπώσει τροπολογίες εξού και οι τέσσερις ε, τροπολογίες των πολιτικών ομάδων αντιπροσωπεύουν 97 σελίδες. Δηλαδή 30-35 σελίδες κάθε τροπολογία και θα χρειαστεί να συγκρίνουμε όλες αυτές τις προτάσεις και να δούμε εάν υπάρχουν ε, διαφορές μεταξύ αυτών που διατυπώνουν η μεν και η δε. Και ήδη την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθώ με τους σκιώδεις εισηγητές και ελπίζω ότι στη συνέχεια θα μπορέσουμε να μελετήσουμε τα προβλήματα που τίθενται και τις ε, ε, διαφοροποίησεις που θα γίνουν και περιμένουν την ε, άποψη των συναδέλφων. Ο κύριος Και εγώ συμφωνώ, πρόεδρε. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια και να κλείσουν όσο γίνεται περισσότερες συμβαστικές τροπολογίες, γιατί είναι το θέμα σημαντικό. Και θεωρώ ότι να δούμε τι θέλει ο συγητής. Γιατί θα πρέπει να είναι σαφές, αποφασιστικό το μήνυμα της Επιτροπής μας για κάποια συγκεκριμένα θέματα, για κάποιες κόκκινες γραμμές ε, διατρέχουμε σημαντικούς κινδύνους τη σημερινή μέρα. Τουλάχιστον όσον αφορά τα θέματα τα δικά μας πρώτα-πρώτα, τι θα γίνει με τους πόρους. Μια που προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει με τους ανατομέα στόχους, πώς να φροντίσουμε να μην ναυαγίσει η πολιτική συνοχής για να πάνε τα χρήματα της συνοχής αλλού, σε άλλες πολιτικές. Με χαρά μου λοιπόν βλέπω ότι είμαστε σύμφωνοι εδώ και δεν θέλουμε να υποκύψουμε στον εκβιασμό. και να θυσιαστούν τα πάντα όπως θέλουν ορισμένοι στην μακροοικονομία. Θα πρέπει επομένω όλοι να δούμε τι, που συμφωνούμε, σε τι, τι, έχουμε κοινά, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι και σε ορισμένα τα θέματα διαφωνούμε και να δούμε τι θα γίνει με αυτό το εν ε, επισυναπτώμενο πλαίσιο ρύθμισης. Έχουμε τις διαφορές μας και με την Περιφερειακή Επιτροπή και με τα όσα λέει ο εισηγητής. Γιατί αυτό το οποίο θέλουμε είναι να είναι αποτελεσματική η πόλη. Να υπάρχει περισσότερος κοινοβουλευτικός έλεγχος. Ε, Επίση να δούμε κατά πόσο θα γίνουν όλα αυτά με κατουξιοδότηση πράξη ή με συναπόφαση. Μέσω του παρατήματος λοιπόν, μέσω ε, των τροπολογιών που έχουμε υποβάλει, θέλουμε να φρενάρουμε την παρακμή του ευρωπαϊκού προτύπου, όλη αυτή την ανεργία στην οποία έχουμε πέσει και το θέμα εδώ, αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο το κοινωνικό ταμείο, είναι όλη, όλη η επιχειρηματική πολιτική. Δεν βλέπουμε τίποτα εδώ να υπάρχει όσον αφορά επομένω τον σημαντικό αυτόν ε, ρόλο, τη σημαντική αυτή προτεραιότητα, το να υπάρχει επομένω ε, ω κοινό ε, παρονομαστή, το πώ θα σώσουμε την απασχόληση, πώ θα τη βοηθήσουμε στην Ένωση. Επίσης, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα τη στρατηγική αυτή. Εμείς έχουμε προτείνει ε, τη σχετική απαλήφη γιατί δεν βοηθάει σε τίποτα. Ε, γιατί εδώ αυτό είναι ο κίνδυνος από αυτά που προτείνει η Κομισιόν. Έχουμε δικαίωμα και οι πολίτες, έχουν δικαίωμα και τα κράτη να ασκούν πολιτική συνοχή. Και αν αντιβαίνει σε αυτό η αποτελεσματικότητα δεν μας λέει τίποτα. Και αλλού έγιναν αυτές οι στρατηγικές. Και δεν ωφέλησαν. Αυτό που, αυτό που πρέπει να αποφύγουμε και αυτό που συνέβη είναι η γραφειοκρατία. Και η οποία γραφειοκρατία δεν αρκεί. Αντίθετα χρειάζεται κάποιο κίνητρο ούτως ώστε κανείς να προχωρεί προ την άσκηση τη ορθία πολιτική γι' αυτό και θέλουμε να γίνουν οι σχετικέ απαλήφες. Επίση, όπω προείπα, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να στείλουμε ένα συγκεκριμένο μήνυμα με τι κόκκινε γραμμέ μα, Ε, γιατί συμφωνούμε καταρχήν ε, και να προσέξουμε να μην υποκύψουμε ε, σε αυτά τα φαντάσματα τα οποία ε, διακρίνουν το πνεύμα των προτάσεων Κομισιών και Κοινοβουλίου. Και επίσης να σας πω το τελευταίο το οποίο με απασχολεί, όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει να γίνει μια αναδιάρθρωση του, των διορθωτικών ε, του, του, του, του Ταμείου Συνοχή, ώστε να καλύψει την ενεργεία των νέων όμως εδώ πέρα κρύβονται κάποιες ε, παγίδες πρώτα πρώτα εάν θέλουμε μια πάγια σταθερή πολιτική ε, τότε θα πρέπει να δούμε το ότι δεν θα πρέπει να είναι προπολογισμό χρόνο με το χρόνο. Χρειάζεται ένα κανονικό ε, κονδύλι. Έτσι θα ωφεληθεί η ανεργία των ε, νέων ή τα μέτρα της ανεργίας. Και επομένως ε, αυτό το οποίο μας λένε είναι ένα καινούριο πρόγραμμα και ότι θα τελικά λένε θα πρέπει να γίνει συρρήκνωση αυτής της πολιτικής στα πάει στο περιθώριο του προπολογισμού. Επομένω, αυτό θα πρέπει να το θεωρήσουμε σαν μια πολιτική συνοχή που εμεί θέλουμε δυνατή με, με κόκκινε γραμμέ και έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε του στόχου που έχουμε τάξει. Κυρία Σαχτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κωσό για την εργασία του σε αυτή την έκθεση. Είναι εξαιρετικά σημαντική. εξαρτάται τόσο από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης όσο και από το παράλληλο δικό μας έργο με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Χρειάζεται λοιπόν να παρακολουθούμε αυτό το συντονισμό και τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων ταυτοχρονών εκθέσεων. Ορισμένα σημεία μου φαίνονται εξαιρετικά σημαντικό να αναφερθούν για αυτή την έκθεση. Το πρώτο σημείο που προσπάθησα να υπογραμμίσω με πολλές τροπολογίες είναι η ένταξη των κοινωνικών εταίρων στις πολιτικές ε, που υλοποιούνται. Θεωρώ ότι οι τοπικές πολιτικές και τα τοπικά προγράμματα θα υλοποιηθούν πιο αποτελεσματικά εφόσον ταυτόχρονα έχουμε τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των διαφόρων ε, συνεργαζόμενων οργανισμών σε αυτά τα έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Δεύτερον, ένα θεμελιώδη σημασία σημείο είναι η τήρηση του 25% που εκχωρείται στο Ταμείο Συνοχής, από το Ταμείο Συνοχής στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Θα πρέπει όλοι μας να συμφωνήσουμε σε αυτό διαφορετικά οι κοινωνικές πολιτικές και είδα άλλη μια απόδειξη σήμερα κύριε Πρόεδρε οι κοινωνικές πολιτικές όλοι κοιτούν να μας τις φάνε, να τις εντάξουν και στο πλήσιο του ΦΕΝΤΕΡ που μας λένε ορισμένες φορές ότι ένα κομμάτι θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στις, πολιτικές, στις κοινωνικές πολιτικές. Το τρίτο σημείο εξαιρετικά σημαντικό είναι η διοικητική απλούστευση της χρήσης όλων αυτών των κονδυλίων και των ταμείων. Το τέταρτο σημείο για το οποίο θα ήθελα να μιλήσω είναι ότι δεν πρέπει απλά να αναφέρουμε τις ε, πολιτικές παιδείας, την αναγνώριση ικανοτήτων, πρέπει να υπογραμμίσουμε και την αναγκαιότητα επαγγελματικής κατάρτασης, για την καλή εκτέλεση και λειτουργία του συνόλου αυτών των προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Κώσα, πρέπει να σας πω ότι είμαι απολύτω στη διάθεσή σας ώστε να συνεχίζουμε να ε, διοργανώνουμε τη διάρθρωση, τη σχέση μεταξύ της δικής σας έκθεσης και της δικής μου έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Κίνγκα Ευχαριστώ. Είμαι πολύ ευγνώμων για αυτή τη συζήτηση, γιατί για μας θα είναι πολύ βασικό το θέμα του κανονισμού αυτού και γι' αυτό χαίρομαι που η κυρία Μπλονσάρ το ανέφερε. Ε, Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να τονίσουμε ότι το, η ελάχιστη συνδρομή του Ταμείου Συνοχής είναι 25% και από εκεί και πέρα κυμαίνεται ανάλογα με το επίπεδο της περιοχής και αυτό θα είναι ένα από τα θέματα κλειδιά. Παρακαλώ λοιπόν επ' αυτού να είμαστε αυστηροί με τις άλλες επιτροπές διότι ξέρω ότι η οι κυβερνήσεις ε, αρέσκονται στο να υπάρχουν ε, τεράστια προγράμματα υποδρομής γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να δαπανηθούν χρήματα σε μεγάλα προγράμματα παιδεία, υποδομή σε άτομα που δεν είναι στην αγορά εργασίας και θα υπάρξει μεγάλη πίεση από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να διηλήσουν την πρότασή μας εξού και θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων, ε, υπάρχει δηλαδή μερική ήδη, ε, ώστε να επιμείνουμε και να μην εγκαταλείψουμε το πρόγραμμά μας. Κάτι άλλο. Το άλλο θέμα που μας ενδιαφέρει είναι ε, η ερεσιμότητα, διότι το συμβόλαιο το Συμβούλιο είπε ότι δεν γίνεται σωστή χρήση των πόρων και ε, εάν κοιτάξουμε την εκ των υστέρων θα δούμε εάν η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί στον ε, επόμενο πρόγραμμα. Εν τω μεταξύ όμως μας ζητούν μία απλοποίηση της διαχειρίσεως των ταμείων αυτών από την βάση, δηλαδή για τις οργανώσεις οι οποίες διαχειρίζονται ε, τα ταμεία αυτά και τους πόρους, να υπάρχει δηλαδή μία αιρεσιμότητα εκ των προτέρων ε, και ε, πρέπει εδώ να πω ότι ορισμένα σημεία τονίζονται και άλλα όχι. Δηλαδή σε ορισμένες περιοχές, σε ορισμένες χώρες ε, η φτώχεια συγκεντρώνεται πολύ περισσότερο στις πόλεις αλλού στην Ήπεθρο και έτσι θα πρέπει να είμαστε ε, ισοσκελισμένοι και να κοιτάξουμε να αναφερόμαστε στα ολοκληρωμένα προγράμματα προγράμματα για την χρηματοδότηση η οποία προέρχεται από διάφορα ταμεία οπότε ε, γι' αυτό και εγώ θα ήθελα εδώ να αναφερθώ στο ελάχιστο ποσοστό του ESF. Το άλλο το οποίο αναφέρεται στον κανονισμό αυτό είναι η αποφυγή των ε, ε, αποκλεισμών που τώρα εμφανίζεται στον κανονισμό αυτό αλλά εάν δεν τονιστεί ενδέχεται στο μέλλον να χαθεί. Γι' αυτό πρέπει να δούμε τους δίκτυες, πόσο θέλουμε να παρακολουθήσουμε την ε, φτώχεια, ποιοι είναι οι στόχοι του 2020 και πώς συνάδουν με το πρόγραμμα αυτό ε, και πώς μπορούμε να ε, προφυλάξουμε τους πολίτες από τα φαινόμενα αυτά μέσω των κανονισμών. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος που έχει ζητήσει να μιλήσει. Όχι. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για αυτό το άρθρο που θα μας απασχολήσει πολύ. Το άρθρο 84.3 του κειμένου του κυρίου Κόζα αλλά και για το ζήτημα της ε, μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Όσον αφορά τη μακροοικονομική αρισιμότητα, δεν θυμάμαι πια ποιο άρθρο είναι. Στη συζήτηση που είχαμε σήμερα το πρωί με τους δύο εισηγητές ε, της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού, του ε, κύριους Μπέργκερ και Καλφίν, είμαι ιδιαίτερα ανήσυχη διότι βαίνουν με τέτοιο ρυθμό οι διαπραγματεύσει που κάθε επιτροπή προχωράει μόνη τη ε, με τη νομοθετική βάση και μετά θα έχουμε το τεράστιο θέμα των ε, αριθμών, αλλά στις νομοθετικές ε, βάσεις υπάρχουν κρυμμένα σημαντικά πολιτικά ζητήματα για τα οποία θα μπορούσαμε ενδεχομένω όλοι μαζί να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση από μια άλλη επιτροπή. Αναφέρομαι σε αυτό το ζήτημα της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας που από αυτή την άποψη είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αν έχω καταλάβει καλά, η πολιτική ισορροπία εντός της Επιτροπής μας δεν είναι ακριβώς ίδια με αυτήν της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης θα προχωρήσει ε, δεν είμαστε σε αναγκαστική συνεργασία για αυτό το τμήμα. Θα προχωρήσει η Επιτρόπη Περιφερειακής Ανάπτυξης με την γνωμοδότησή της χωρίς οι πολιτικές ομάδες και η και η ε, ολομέλεια να μπορούν να αναφερθούν σε αυτό το ζήτημα. Πιστεύω ότι αυτή εδώ είναι η κατάλληλη στιγμή να θέσουμε το πρόβλημα ώστε ε, ο καθένας, η κάθε πολιτική μας ομάδα να το έχει υπόψη της. Εάν δεν γίνει τίποτα, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως καταλαβαίνω, είναι υπέρ της μακροοικονομικής ερεσιμότητας και αυτό μπορεί να υπερισχύσει και στη συνέχεια για να αλλάξουμε τη θέση του Κοινοβουλίου δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Δεν είδα τη συμβιβαστική τροπολογία που μας προτείνει ο συγκητής για αυτό το σημείο. Εγώ κατάλαβα ότι στην Επιτροπή μας είμαστε οι περισσότεροι κατά αυτής της μακροοικονομικής ερεσιμότητας Σε αυτό το σημείο λοιπόν δεν πρέπει να παραμείνουμε με την απόψή μας κλεισμένοι σε αυτή την αίθουσα, θα πρέπει να επηρεάσουμε και έξω από αυτήν τα πράγματα. Επίσης κάπως επίσης οριζόντια το άρθρο 84 παράγραφος 3 εκεί μπορώ να, μπορώ να είμαι πιο ακριβής γιατί το είχα προβλέψει το ζήτημα είναι να δούμε πόσα θα δεσμεύσουμε για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. για την μετάβαση για αυτές τις τρεις κατηγορίες ε, περιφερειών στις οποίες αναφέρομαι. Εκεί τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Ε, αν δούμε ποιο είναι το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων όπως το έχει προετοιμάσει η Δανική Προεδρία, αυτά τα ποσοστά ήδη έχουν προβληθεί. Και στο πνεύμα της Δανικής Προεδρίας αποτελούν κομμάτι της διαπραγμάτευσης όπως και τα ποσά του δημοσιονομικού πολιτικού πλαισίου το οποίο κατά εμάς είναι απολύτως απαράδεκτο σημαίνει ότι ο καθένας μας πρέπει να κινητοποιήσει τους, ε, την μόνιμη αντιπροσωπεία του ώστε να μην αφήσουμε να γίνει κάτι τέτοιο μεθαύριο στο Συμβούλιο της ΕΠΣΚΟ διότι η ΕΠΣΚΟ θα μελετήσει λίγο το διαπραγματευτικό αντικείμενο αλλά στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου που θα προετοιμάσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και όπου εάν στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ε, το αποτέλεσμα της διαπραγματευσής όπως έχει προετοιμαστεί από τη Δανική Προεδρία εγκριθεί, όλα ξανανοίγουν. Μελετήσαμε και παρακολουθούσαμε αυτό το πρόβλημα από την αρχή στην Επιτροπή μας. Ορισμένοι θα θυμούνται ότι αρχικά ο Επίτροπος και η Γενική Διευθύνση του είχαν, προβλε... είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο το να βγάλουν εντελώ από τα διαρθρωτικά ταμεία το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει μια κοινωνική πολιτική και τα μέσα για να δράσουμε. Ορισμένα μέλη και από την Επιτροπή μας στη συνέχεια έπεισαν ότι έπρεπε όλα να είναι σε ένα, κοινωνικό, σε ένα κοινό πλαίσιο και μετά μπορούμε να κάνουμε θέλουμε. Αυτό το κοινό πλαίσιο είναι υπερβολικά μεγάλο και μέσα σε αυτό το πλαίσιο καταστρέφουμε αυτή τη στιγμή την κοινωνική πολιτική. Σας το τονίζω, εάν δεν ε, ενωτήσουμε, ενοποιήσουμε αυτό τα ποσά, εάν δεν τα σταθεροποιήσουμε, τέλος στην κοινωνική πολιτική. Και όταν βλέπω την κατάσταση σε ορισμένες χώρες, ειδικότερα τις πιο απομακρυσμένες, μην μου λέτε ότι αυτό που χρειάζεται περισσότερο Πορτογαλία σήμερα είναι οδικές υποδομές. Δεν είναι αλήθεια. Υπάρχει εδώ μια ισορροπία διαρθρωτικών πολιτικών όπου αγαπητέ κύριε Σαγητά εσείς είστε ο σημειοφόρος μας. Θα πρέπει να ε, τονίσετε, να επισημάνετε έντονα ορισμένα πράγματα ήδη αυτή την εβδομάδα παρότι πρόκειται για μια ευθύνη την οποία θα πρέπει να φέρουμε όλοι μαζί, μαζί σας. Αυτά είναι τα δύο σημαντικότερα σημεία που ήθελα να αναφέρω σε αυτή τη φάση, χωρίς να επανέλθω σε κάποιες πτυχές ε, για τα υπόλοιπα προς ε, ρεστοποίηση και άλλες πτυχές που ανέφεραν ορισμένοι συνάδελφοι. Θα ήθελε η Κομισιόν να μιλήσει. Oui, non. Oui. Ίσως να πείτε κάτι για τη συζήτηση έτσι όπως ε, έχετε αντιληφθεί ότι λαμβάνει η χώρα στο Συμβούλιο όσον αφορά αυτή την κάμψη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε σχέση με τα Ταμεία Συνοχής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τον ε, ε, εισηγητή για αυτά τα οποία έκανε και το πρόβλημα των πόρων εντάσσεται στην προβληματική για το πολιτές χρηματοδοτικό, δημοσιο... χρηματοδοτικό πλαίσιο, το MFF, και όσον αφορά την εταιρική σχέση, ε, είναι το θέμα οριζόντιο. Για αυτή την εταιρική σχέση, πολλοί βουλευτέ εκφράστηκαν σε σχέση με αυτή την εταιρική σχέση για την οποία εμείς θέλουμε, αν θέλουμε να, να, να, να έχει ποιότητα θα πρέπει μόνο έτσι να εξυπηρετεί τις περιφέρειε ένωσης. Ο δε κώδικας διοντολογίας είναι πάρα πολύ βασικό εργαλείο τόσο ώστε να ωφεληθούμε από αυτή την εταιρική σχέση. Όσον αφορά τώρα το πλαίσιο της ε, το, απόδοσης, και εμεί θεωρούμε ότι χρειάζεται μακροοικονομική αιρεσιμότητα και όπως γνωρίζετε, αυτό το πλαίσιο απόδοσης το θέλουμε για να υπάρχουν επιπτώσεις θετικές από τους πόρους. Αν κλαδέψουμε τις φιλοδοξίες μας, δεν θα ωφελήσει όσον αφορά την τοποθετικότητά μας να είναι αποδοτικά τα προγράμματα και άρα πρέπει να συζητήσουμε κάποιες βελτιώσεις ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα των προγραμμάτων. Τώρα όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων και την αποφυγή των διακρίσεων, ευχαριστούμε για τις προσπάθειες βελτίωσης της προτάσεώς μας. Είμαστε στη διάθεσή σας για να τα συζητήσουμε. Και έτσι όλα αυτά να τα εφαρμόσουμε στην καθημερινή άσκηση της πολιτικής συνοχής. Bon, euh, monsieur, je vais être Αγαπητέ κύριε, θα είμαι δυσάρεστη. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά, μου συμβαίνει. Ειλικρινά, όταν η Κομισιόν έρχεται να μιλήσει εδώ για να ευχαριστήσει τους βουλευτές για τη συμβολή τους, είστε εκτός θέματος. Βρισκόμαστε ενώπιον ενό μιας νομοθετικής πρότασης την οποία γράφουν οι βουλευτές. Είμαστε συνομοθέτε. Σταματήστε λοιπόν να έρχεστε από την Κομισιόν και να μας λέτε που είστε πολύ χαρούμενοι με τις τροπολογίε σας. Δεν μας ενδιαφέρει. Έχουμε δικαίωμα πρωτοβουλίας, έχουμε δικαίωμα ως νομοθέτε. Τέλο. Ζητώ συγγνώμη. Ήθελα να το πω εδώ και πολύ καιρό και το λέω τώρα. Και μάλιστα δεν το έκανα, δεν το είπα σήμερα το πρωί. Θα επανέλθω σε ένα σημείο και θα σας ξαναδώσω τον λόγο. Όσον αφορά το σχόλιο τεχνικής φύσης που κάνατε, όσον αφορά το ρόλο της Κομισιόν της εργασίας μας, όσον αφορά το, στρατηγικό κοινό, το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, όσον αφορά το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, πώς βλέπετε τα πράγματα διότι θα αντιληφθήκατε ότι υποβλήθηκαν τέσσερις τροπολογίες οι οποίες καλύπτουν το σύνολο του εγγράφου και εμείς ε, βρισκόμαστε σε αβεβαιότητα, δεν ξέρουμε τι θα κάνει η Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων, θα τα εντάξει στο πλαίσιο της συναπόφασης, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα που εσείς διακρίνετε σε αυτό το κείμενο όπως θα εξελιχθεί. Γνωρίζετε ίσως ότι έγιναν συζητήσεις για να δούμε κατά πόσο πρέπει να κρατήσουμε αυτό το έγγραφο εκτός της, της συναπόφασης ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία. Ταυτόχρονα εφόσον ενταχθεί στη συναπόφαση θα θέλαμε να είμαστε και εμείς μέλος διαπραγμάτευσης. Πώς βλέπετε την κατάσταση αυτού του εγγράφου ουσιαστικά σας δίνω την ευκαιρία να επιχειρηματολογήσετε υπέρ της λύσης που εσείς παρουσιάσατε. Αλλά θεωρώ ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου θα, χρειαστεί, θα χρειαστούν περισσότερες διευκρινήσεις. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Κομισιόν είχε προτείνει το κοινό στρατηγικό πλαίσιο να εγκριθεί με κατεξοδότηση πράξη οι διάφορες προτάσεις που έγιναν και στην Επιτροπή Απασχόλησης είναι το να είναι παράρτημα του κανονισμού η Κομισιόν μπορεί να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο με αυτή, σε αυτή τη βάση. Να συμπεριλάβει το μηχανισμό συντονισμού και το μηχανισμό συνοχής στις υπόλοιπες ενωσιακές πολιτικές ως παράρτημα του κανονισμού. Αντιθέτως, οι δράσεις κλειδί, οι πρωταρχικές κύριες δράσεις, ε, οι εδαφικές προκλήσεις και οι τομείς προτεραιότητας όσον αφορά τη συνεργασία θα ε, αποτελέσει το αντικείμενο μιας ξεχωριστής κατεξουδότησης πράξης. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ελπίζω ότι αυτό θα επιτρέψει να απαντηθούν οι ερωτήσεις σας. Τι βάζετε στις κατεξουδότησης πράξεις στην το κομμάτι που θα τοποθετηθεί ως παράρτημα στον κανονισμό θα είναι η επιλογή πολιτικής, ο μηχανισμός συντονισμού και ο μηχανισμός που ε, διασφαλίζει τη συνοχή με τις υπόλοιπες πολιτικές. Όλα αυτά θα προσαρτηθούν στον κανονισμό. Αντιθέτως, οι δράσεις κλειδιά, οι δράσεις προτεραιότητας, οι εδαφικές ε, προκλήσεις και οι τομείς προτεραιότητας για τις δραστηριότητες συνεργασίας θα αποτελέσουν το αντικείμενο ξεχωριστής κατεξουσιοδότηση πράξη. Αυτή είναι σήμερα η πρόταση της Κομισιόν, έτσι λέτε. Ναι, απολύτως. Κύριε Ισηγητά, δεν ξέρω αν θέλετε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Κώστα. Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμο αυτό το οποίο άκουσα. οι συνάδελφοι είπαν πράγματα με τα οποία όσοι τουλάχιστον συμφωνώ. Άλλωστε δεν είναι συμπτωματικό τότε συμφωνήσαμε και με τους σιώδης ηγητές την περσμένη εβδομάδα. Όπως είπε η κυρία Πρόεδρος, μπορούμε μαζί να προχωρήσουμε. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε έτσι την ε, αποκρισταλωμένη θέση της Επιτροπής Απασχόλησης. Πάντως ε, υπάρχει κάτι εδώ που δεν μου αρέσει. Ότι δηλαδή μίλησαν μόνο οι βουλευτές του Λαϊκού Κόμματος και του Σοσιαλιστικού. Οι άλλες πολιτικές ομάδες το πιο σωστό είναι να υπάρχει ευρεία συνένεση. Επομένω, εγώ θα πάω να αναζητήσω τη γνώμη των άλλων πολιτικών ομάδων και θα περιλάβω και την δική τους θέση στην γνωμοδοτησή μου. Τώρα, έχω εγώ τρεις συγκεκριμένε ερωτήσεις. Πρώτον, ήδη είχαμε μια δεύτερη εκδοχή της ε, εκθεσιός μου. Θεωρούμε ότι η συναπόφαση είναι μια διαδικασία πολύ σημαντική. Οπότε αυτό ριοθετεί και την αρμοδιότητα της Κομισιόν να ενεργεί με βάση κατεξοδότηση πράξης. Αυτό το οποίο να γίνει είναι το 25% να συνεχίσει να ισχύει και ακριβώ έτσι είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι. Άρα δεν νομίζω ότι εδώ πέρα θα έχουμε πρόβλημα. Και αυτό αφορά και το πώς θα καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τώρα για τις τροπολογίες, ήδη έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο αποσκοπεί στο να μειωθεί η γραφειοκρατία. Θα πρέπει να διευκολυνθεί από ε, όλη, όλη η, η διαδικασία. Πάντως ούτε είναι τόσο σίγουρο ότι οι πολίτες, οι μισθωτοί, οι περιθωριοποιημένοι θα συμφωνήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω θα υπάρξει αντιπαράθεση. Πάντω. θα ήθελα οι συνάδελφοι να σκεφτούν το εξή. Θα ήθελα να συμφωνήσουν με τι συμβαστικέ που κλείσαμε με τους χιώδες ηγητέ. Και συμφωνώ ότι θα πρέπει όλοι μας, ο καθένας στην πολιτική του ομάδα, να προωθήσει αυτά που θα συμφωνήσουμε. Όταν εξηγηθεί για τρίτη φορά αυτό το κείμενο, νομίζω ότι τότε θα μπορέσουμε να κλείσουμε συμβασμό σωστό. Πολύ ωραία. Ακούστε κύριε Σιγητά, σας εύχομαι λοιπόν καλό κουράγιο και ελπίζω ότι με τους κοιόδης συζητητές θα καταφέρετε να καταλήξετε σε ικανοποιητικούς συμβιβασμούς τους οποίους θα πρέπει να υιοθετήσουμε έως τις 5 Ιουλίου. Κάνω λοιπόν την ίδια παρατήρηση και για την κυρία Μόρα αρχίσει σήμερα το πρωί. Πιστεύω ότι για το σύνολο των συναδέλφων είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στη διάθεσή μας την επόμενη εβδομάδα συμβιβαστικές... Ξέρω ότι έχετε στείλει στις τις συμβιβαστικές σας τους συναδέλφους. Αλλά τώρα έχετε να εργαστείτε με τους Κιώδης και να διορθώσετε αυτές τις συμβιβαστικές βάσει των συζητήσεών σας με τους Κιώδης. Θα πρέπει λοιπόν και τα υπόλοιπα μέλη να ε, μάθουν ποια είναι η τελική, σε τι συμφωνήσει τελικά. Πριν από την ψηφοφορία της 5ης Ιουλίου στο Στρασβούργο. Περνάμε στο σημείο 15 της ημερήσιας διάταξης και δίνω τον λόγο στον κύριο Μπέκερ για να συζητήσουμε τις δια... 83 τροπολογίες για την πρωτοβουλία του για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την πρόθεση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, σας πω καταρχήν πού βρίσκονται οι εργασίες σχετικά με την έκθεση αυτή και να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής για την πολύ ενεργή συμμετοχή όχι μόνο των σκιωδών εισηγητών αλλά και των συντονιστών της πολιτικής ομάδος και των ε, βοηθών στην ομάδα μου. Μπορώ να σας πω ήδη ότι ο μεγάλος αριθμός των τροπολογιών ε, απλά από πλευράς αριθμού και από περιεχόμενο αντικατοπτρίζουν τη σημασία αυτού του θέματος διότι πρέπει να πούμε ότι η έκθεση για τις, ε, την κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ένα ενδιαφέρον θέμα και λαμβάνει χώρα σε μια πολύ επίκαιρη στιγμή διότι υπάρχουν πολλά περιεχόμενα τα οποία περιέχονται σε άλλες εκθέσεις όπως το Κοινωνικό Επενδυτικό Ταμείο ή την έκθεση Στάινμπρουκ ή στην έκθεση Ο Κορνέ που αναφέρονται σε παρεμφερή θέματα. Υπάρχουν δηλαδή διατάξεις οι οποίες ε, λαμβάνουν χώρα κατά κάποια στιγμή ε, χρονική που προ καταλαμβάνει ήδη τη δικιά μας έκθεση. Εξού και κάθε έγγραφο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει από διαφορετική σκοπιά το κείμενο. Είτε πρόκειται για τα αγγλικά, είτε πρόκειται για τα γερμανικά, είτε για κάποια άλλη γλώσσα. Δηλαδή ε, αυτή τη στιγμή ε, πολύ απλά και πολύ συνειδητά θέλω να πω ότι είναι γεγονός και πρέπει να το παραδεχθούμε ότι αυτό το οποίο προσπαθώ εγώ δηλαδή την όλη θεματολογία να την ε, αντιμετωπίσω σε συγχρονισμένα κατά τρόπον ώστε να έχουμε ακριβείς ορισμούς και στο μέλλον ε, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους κοινωνικούς ε, επιχειρηματίες. Τι είναι τα θέματά μας, ουσιαστικά τρία. Δύο θέματα κλειδιά που ε, ο καθένας βλέπει από διαφορετική οπτική γωνία, η επανεπένδυση και η συμμετοχική ε, συνδρομή. Προσπαθώ λοιπόν όσον αφορά την καινοτομία, όσον αφορά τις νέες εξελίξεις οι οποίες ε, ξεκινούν από την αλλαγή των συνθήκων που ε, προέκυψαν εφέτος και θα μας ανοίξουν νέες δυνατότητες, αυτές τις δυνατότητες να τις προωθήσω και να μην τις εμποδίσω, αντιθέτως να τις προωθήσω και να τις διατυπώσω πιο σαφώς. Αυτή είναι η σκέψη ε, βάση της οποίας προχωρώ και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική. Πέραν αυτού υπάρχει και μία ευθύνη εκ μέρους μας, δηλαδή οι μελλοντικέ δυνατότητες θα πρέπει να καταστούν δυνατές και να βοηθηθούν με κάθε τρόπο και με μέσα. Εξού και οι τροπολογίες θα μπορέσουν να βοηθήσουν στη διευκρίνηση του κειμένου και το τρίτο κριτήριο είναι ε, αυτό το οποίο ε, ε, εξασφαλίζει ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα πρέπει να έχει ένα, μια κοινωνική επίπτωση, μια κοινωνική αποτελεσματικότητα και αυτό θέλουμε να τονίσουμε. Προσπαθώ να σας πω ότι στο χρόνο που έχουμε ε, των επομένων 15 ημερών ε, ε, θα συναντηθούμε με τους σκιώδες και θα προσπαθήσουμε ως το δυνατόν πιο γρήγορα να σας υποβάλουμε μαζί με τους σκιώδεις εισηγητές κείμενα κατά τρόπον ώστε να διερευνήσουμε και να εξεύρουμε εντός δύο εβδομάδων τις εναλλατικέ λύσεις που θα καταλήξουν σε ένα κείμενο που θα τύχει ευρείας αποδοχής. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει η κυρία Να επαναλάβουμε αυτά που είπε στην αρχή του ο εισηγητής είναι εκθεσιτία πρωτοβουλία αλλά το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Και αυτό αποδεικνύεται από όλε αυτέ τι τροπολογίε που έχουν υποβληθεί. Και εγώ επομένω θεωρώ ότι θα είναι τιτάνιο το έργο να εξεταστούν όλε αυτέ. Πάντω, βλέπω κάποιε γενικέ αρχέ, γενικέ κατευθύνσει που τι διέπουν και νομίζω ότι θα πρέπει η Κομίσιο να βοηθήσει να εξασφαλίσουμε κάποιο επίπεδο νομικό ε, και οικονομικό που να βοηθήσουν έτσι τους ενδιαφερόμενους. και τους ορισμούς, κοινωνικές οικονομίες, κοινωνικών επιχειρήσεων και όλα αυτά κάπως να αλληλοσυνδεθούν για να προσθέσουμε κάτι στα όσα ήδη έχουμε καταλήξει ως θέση ως μήνυμα. Να δούμε πώς θα βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση των κοινωνικών επιχειρήσεων. Όλοι από ό,τι φαίνεται συμφωνούν ότι το κοινωνικό επιχειρήν βοηθά πάρα πολύ στο να απαλληλθούν οι επιπτώσεις της κρίσης. Επίσης, δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Και επομένως, αυτό που θέλουμε είναι να εξετάσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Με όσο βλέπω, θα κάτσουμε και θα, να προσέξουμε να μην καταρρεύσει η έκθεση από τις τόσες τροπολογίες. Πάντως, είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Μπέκερ κάτι θα βρει για να βοηθήσει σε αυτό που έχουμε όλοι σαν κοινό σκοπό. Πώς θέλει Πρόεδρος, θέλει όλος το λόγο. Ε, για λογαριασμό του Σβέν σας μιλώ. Θεωρούμε ότι θα πρέπει αυτή η έκθεση να στηριχθεί περισσότερο σε όσα ήδη έχει κάνει το Κοινοβουλίο. Όπως ας πούμε η έκθεση του Σβέν. Να μην υιοθετήσουμε νέους ορισμούς, λέει κύριε Τούρν. Συμφωνία με των πολιτικών ομάδων και επ' αυτού να στηριχθούμε και να προχωρήσουμε. Επίσης, πρόσβαση σε πιστώσεις και χρηματοδότηση. Πολύ σημαντικό αυτέ τι επιχειρήσει. Η διασύνδεση με την στρατηγική του 2020 και εδώ και τους ορισμούς. και κοινωνική επιχείρηση. Να προσέξουμε επομένως γιατί κανείς έτσι κινδυνεύει να δημιουργήσει μια μεγάλη γκρίζα φαιά περιοχή όσον αφορά την εταιρική ευθύνη των ε, κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων. Και θα έχουμε και κάποιες τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Να πω και εγώ δύο λόγια. Γιατί όλοι χαίρονται μια έκθεση για πρωτοβουλίε για ένα τέτοιο θέμα που μα είναι τόσο αγαπητό. Όμως υπάρχει εδώ πέρα μια μεγάλη δυσκολία. Επί τραπέζι βρίσκεται αυτή η έκθεση. Και τελικά θα πρέπει να δούμε γιατί αυτή η έκθεση την εξετάζουμε παράλληλα με άλλες, άλλες πρωτοβουλίες που έχουν ολοκληρωθεί ή όχι. Αναφέρθηκε το σχετικό με τους αλλά έχω και άλλες δύο πρωτοβουλίες. Την έκθεση Όκονη στην Οικονομική Νομισματική Επιτροπή. Θα κάνουμε εκεί κάτι όσον αφορά την ε, κοινωνική εταιρική σχέση, την κοινωνική συνεργασία. Και από την άλλη μεριά έχουμε την έκθεση της Γιούτα όσον αφορά την ε, την ε, καινοτομία, οπότε θα προσπαθήσουμε, εν να καλύψουμε τις ε, προτάσεις του κυρίου Μπέικερ. Τώρα, τι να σας πω, δεν είναι δικός μου ρόλος, αλλά το λέω ως μέλος της Επιτροπής, ότι θα πρέπει να καταβάλει διετή προσπάθεια ο εισηγητή πρωτα Πρώτα-πρώτα, να δει το ότι Ωραία, σε όλους μας αρέσουν αυτές οι θέσεις της πρωτοβουλίας, αλλά για να μην απλή φιλολογία θα πρέπει να προσέξουμε. Θα πρέπει κάπου να καταλήγει, αλλιώ είναι ε, μεγάλη απογοήτευση η πολιτική που δεν καταλήγει να πω. Για να δούμε ποιο ακριβώ είναι το μηχάνημα. Το, συγγνώμη, το μήνυμα το οποίο θέλουμε να στείλουμε αυτή την έκθεση. Ποια είναι τα, τα, τα δύο-τρία πιο σημαντικά στοιχεία κλειδιά και πώ θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε το ότι θα ε, είμαστε συνεπείς με τα όσα ήδη έχουμε κάνει. Δεν είναι το, το, το, το, το κοινωνικό επιχειρήν, α πούμε. Έτσι θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπαθίες μας για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάτι από όλες αυτές τις τροπολογίες που δεν είχα ούτε το χρόνο ούτε το θάρρος να τις διαβάσω. Αυτά ήθελα κύριε εισηγητά. Πάντως, αυτό που όλοι θέλουμε είναι αυτή η έκθεση να είναι όσο γίνεται πιο αποτελεσματική. Ο Σίγητς έχει το λόγο, μια που άλλο το λόγο. Μπέκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι ουσιαστικά στην αρχή ε, είπα ότι αυτό που μας απασχολεί είναι το θέμα των ορισμών, της ορολογίας που είναι ένα δύσκολο έργο διότι υπάρχουν διαφορετικοί διαφορετικής ε, χρησιμοποίησης όρων αναλόγως των ε, εγγράφων και πρέπει να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε όλο αυτό το εύρος. Επίσης, συμφωνώ απολύτως ότι θα πρέπει να δούμε και την ε, οικονομική βάση για το κοινωνικό επιχειρήν και να δούμε από ποιες πηγές μπορεί να προέλθει. Πρέπει να διαρθρωθεί η έκθεση επιπλέον, δηλαδή βάσει των τροπολογιών θα ακολουθήσουμε την ε, σειρά των ε, κεφαλαίων και θα την καταστήσουμε πιο ορθολογική. Ε, κύριε Κίγολτ, θα ήθελα να σας πω ότι ακριβώς το γεγονός ότι βασιζόμαστε σε εργασίες οι οποίες έχουν ήδη γίνει είναι ένας από τους λόγους γιατί πρέπει να ε, ε, αντιταχθούμε σε ορισμένες απόψεις επί των οποίων υπάρχουν ε, ήδη γραπτά. Και Όσον αφορά τον προσανατολισμό προς το κέρδος ή όχι, όπως είπα στην αρχή ρητός, ε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί συζήτηση και πρέπει ρητός να σας πω ότι εγώ προσωπικά είμαι της απο, αποψής ε, και έτσι ε, θα προβώ και σε συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές ότι πρέπει να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για νέες με συνεργασίες. Και ε, μπορώ να σας πω ότι η, η Αυστριακή ε, Οργάνωση Καριτάς έχει μία 100% φυγατρική εμπορική της Καριτάς που είναι θρησκευτική οργάνωση η οποία ε, ε, λέει στο καταστατικό της ότι πάση θυσία πρέπει να υπάρχουν κέρδη και αυτό από μια οργάνωση η οποία επιζητεί κοινωνικούς στόχους. Αυτό σας δείχνει ότι υπάρχουν και κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες θα χαρούν πάρα πολύ εάν υπάρξει ε, εάν ε, ε, ε, τις απαγορεύσουμε τις, τα ρητά κέρδη παρόλο που δεν θα τις βοηθήσουμε. Εμείς όμως δεν θέλουμε να καταστήλουμε τις δραστηριότητες, θέλουμε να δημιουργήσουμε καλύτερες προοπτικές. Κυρία Πρόεδρε, με αυτά που είπατε μου μιλάτε πραγματικά, με πιάντε στο συνέστημα, διότι όπως σας είπα πάρα πολύ σαφώς θεωρώ ότι η εργασία εργασία της κυρίας Στάινμπρουκ ενσωματώθηκε ε, ε, ε, συνειδητά στην δικιά μου εργασία κατά τρόπον ώστε ο συγχρονισμός των δύο αυτών εκθέσεων οδηγήσει σε έναν πιο συνεκτικό στόχο και θα ήθελα το θέμα αυτό να απασχολήσει και τους σκιώδεις εισηγητές. Δηλαδή ε, δεν θέλω εκ προημίου να προκαταλάβω πώς θα πρέπει να λειτουργήσουμε αλλά πιστεύω ότι λόγω του ε, υψηλού αριθμού των τροπολογιών θα χρειαστεί τις ε, επόμενες ημέρες να συνεργαστούμε με τους σκιώδεις εισηγητές και πιστεύω ότι είμαστε σε σωστό δρόμο. Πολύ ωραία. Αφού έχουν έτσι λοιπόν τα πράγματα... Είναι 10 Ιουλίου, όχι αυτή είναι μια άλλη συνεδρίαση. Ε, θα εξετάσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες σας στις 10 Ιουλίου και νόμιζα για μια στιγμή ότι ήταν 5 Ιουλίου που ήδη είναι μια μέρα με πολλά θέματα στην ημερησία διάταξη. Περνάμε στο σημείο 16. Δίνω τον λόγο στον Αλεχάνδρο Σέρκας για την παρουσίαση της έκθεσης πρωτοβουλίας του για την ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζόμενους, πρόβλεψη και διαχείριση της αναδιάρθρωσης. Κύριε Ισηγητά, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα θα αρχίσει μια μακρά διαδρομή η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί με μια σύσταση για να έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο ή θα πέσει στο κενό και όλα θα συνεχίσουν όπως είχαμε πριν. Περί πρόκειται, περί πολύ σημαντικού θέματος για την σημερινή και για την ε, αυριανή Ευρώπη. Μιλάμε για τις αναδιαρθρώσεις, τις μετακαταστάσεις, τεχνολογική αλλαγή, το μέλλον της βιομηχανίας. Μιλούμε για τους πυλώνες, τα βασικότερα κεφάλαια επί των οποίων φτιάχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ΕΚΑΦ αρχή. Μεγάλο πρόβλημα και μεγάλη ευκαιρία για να διαρθρώσεις. Πάντοτε ήταν κάτι το εγγενές για την βιομηχανική επανάσταση, την τεχνολογική αλλαγή, την καινοτομία, την αλλαγή. Είναι πάρα πολύ βασικό ότι όταν δούμε τα αριθμητικά στοιχεία η κατάσταση χαρακτηρίζεται σαν μια συνεχής τραγωδία. Εδώ και τέσσερα χρόνια έχουμε κρίση που μαστίζει την ε, βιομηχανία και μόνο 4.000 αναδιαρθρώσεις σύμφωνα με το παρατηρητήριο του Δουβλίνου Έχουμε χάσει λοιπόν λόγω αυτών των διαρθρώσεων, μάλλον παρά αυτές των διαρθρώσεων, έχουμε χάσει 1.800.000 θέσεις εργασίας. Τη βιομηχανία δουλεύει μόνο ένα στους εξεργαζομένους. Είναι το να ζήσουμε μόνο από, την, ε, από τις υπηρεσίες, δεν γίνεται χωρίς την ε, ε βιομηχανία. Πρόκειται για μια πρόκληση πρόκειται για μια ευκαιρία. Χτες συνάντησα εργαζόμενους από την Αρσελόρ. Και λέγανε ότι χάθηκαν 30.000 θέσεις εργασίας, έτσι του έτσι απειλείται ε, και ενώ το αρμόδιο αρμόδιο υπηρεσία είναι στο Λουξεμβούργο, ουσιαστικά οι, απο, αποφάσεις λαμβάνονται στο Λονδίνο. Σαν επομένως να ήταν θέμα ε, επιχείρησης μόνο και όχι θέμα της κοινωνίας, σαν να ήταν θέμα μόνο των μετόχων. Ενώ τελικά ε, το θέμα είναι θέμα όλες τις, τις περιφέρειες που, που μένουν οι εργαζόμενοι. να σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι αυτά θα αυτορυθμιστούν ε, μόνο επί τη βάση των συμφερόντων των ε, μετόχων. Στις 28 Ιουνίου η Όπελ θα λάβει πάρα πολύ σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον τη. Να δούμε τι θα γίνουν όλα αυτά τα εργοστάσια. Τι είναι, είναι θέμα μετόχων, είναι θέμα κοινωνίας, θέμα πολιτικής, θέμα των εκπροσώπων κοινωνία. Να, ποια είναι η προβληματική συνάδελφη δεν είναι θέμα μόνο μιας χώρας ή μόνο ενός κόμματος. Είναι κάτι που αφορά όλη την Ευρώπη και η ένταση είναι πρωτοφανής. Δεν είναι δυνατόν τα χρηματιστήρια να κατησχύουν της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας. Θα πρέπει να περτανεύει ο κοινωνικός διάλογος γιατί η κρίση έφερε μια πίκρα και ξεχάσαμε ότι είμαστε κοινωνία που θέλει να είναι ανταγωνιστική. Η οικονομία της αγοράς, αλλά μπορεί να είναι ανταγωνιστική, αλλά δεν θα πρέπει ποτέ όλα αυτά, αυτές οι φιλοδοξίες, να βάζουν στην άκρη τις υπευθυνότητές μας, τις ευθύνες μας σε σχέση με τους εργαζομένους. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, αναδιαρθρώσεις σωστές και αναδιαρθρώσεις που έγιναν λάθος. Οι σωστές δίνουν ευκαιρία σε περιφέρειες, σε επιχειρήσεις, σε κράτη και σε εργαζομένους. Ξέρουμε τι γίνεται όμως με αυτές που δεν πάνε καλά και ξέρουμε πώς γίνονται οι καλές και πώς γίνονται και οι κακές που είναι η πλειοψηφία. Εγώ έχω εδώ στην είσοδο ένα έγγραφο. Στο έγγραφο αυτό αναφέρονται κάποιες ε, μελέτες που έχουν κάνει πανεπιστήμια σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα και βλέπουμε πού είναι τα λάθη. Βλέπουμε ποιες πετύχαμε, ποιες πετύχαμε και ποιες απέτυχαν. απέτυχαν. Γιατί απέτυχαν, απέτυχε η πλειοψηφία, γιατί δεν έχουμε μέσα, ούτω ώστε με τρόπο οριζόντιο και υποχρεωτικό, να κάνουμε αυτές τις αναδιορθώσεις να, αυτές υπόψη υποχρεωτικά τις άριστες πρακτικές. Είχε πριν από λίγο καιρό μια πράσινη βίβλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν από 10 χρόνια γίνονταν σεμινάρια, αναλύσει, ερωτήσει και όλα τελικά φέθηκαν στην καλή πίστη, στην καλή διάθεση. Υπάρχουν κάποιε χώρε που ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρόκληση, υπάρχουν κάποιε εταιρείε που το κάνανε αυτό. Μα δίνουν παράδειγμα, αλλά υπάρχουν άλλε οι οποίε δεν, δεν ε, αντέδρασαν. Οπότε, η προ, το πρώτο κομμάτι τη εκθέση μου, εκεί δικαιολογώ το γιατί πρέπει να αναλυθεί δράση. Ε, γιατί πρέπει κάτι να γίνει στην ιστορία της Ευρώπης που τώρα στη σημερινή συγκυρία έχουμε ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό. Ένα ευρωπαϊκό που θα πρέπει να αποφασίσουμε τη μεθοδολογία να το επιλύσουμε. Τι θέλουμε. Νομοθεσία ή ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό το οποίο να υποχρεώνει τη λήψη υπόψη των αρίστων πρακτικών και την εμπλοκή όλων των ε, κοινωνικών εταίρων αν το θέλουμε αυτό μπορεί να γίνει. Και αφού πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει, γιατί να μην το κάνουμε. Γιατί να, μην, σταματήσουμε την, ε, την, ε, το, να πληγώνεται της Ευρώπη να φιλορροεί. Όχι, δεν μπορεί και αυτό να αυτορυθμιστεί μόνο, δεν μπορεί να το κάνει αυτό μόνο, του, μόνο, του, μόνο της η αγορά. Η αγορά προσέχει τους μετόχους. Ο κύριος Μιτάλ είναι ε, κάτι σαν αρπακτικό και αν η Ευρώπη δεν βασίζει τα φέροντά τη, τότε θα βγει χαμένη. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, κάτι να κάνουμε. Το δεύτερο τμήμα τώρα είναι το τι μπορούμε να κάνουμε. Οδηγία. Οδηγία πλαίσιο η οποία σε αυτά τα πλαίσια να θέτει τα, τα, τα ελάχιστα, τις ελάχιστες τα οποία, αν δεν υπάρχει ανταπόκριση από το κράτος, να ενεργοποιούνται αυτά τα ελάχιστα. Σε περίπτωση που δεν έχουν συμφωνήσει οι κοινωνικοί εταίροι. Εκεί που πάνε να εφαρμόσουν αυτό το, το, το, το απίστευτο, το να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. αυστηρό παιδί εφαρμογή, καλά περιχαρακωμένο, καλά καθορισμένο. Όσον αφορά τους ομιλου επιχειρήσεων, τις μεγάλες επιχειρήσει που αναδιαρθρώνονται και τις θηγατρικέ. Για τις σημαντικέ, τις μεγάλες αναδιαρθρώσεις εκεί που έχουμε πάνω από 100 εργαζομένους. Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε με τίποτε παραπάνω της ΜΜΕ. Δεν θέλουμε να τους κάνουμε τη ζωή πιο δύσκολη, θέλουμε να τις βοηθήσουμε. Ούτως ώστε να πετυχαίνουν οι αναδιαρθρώσει οι σωστέ είναι αυτέ που έγιναν επί τη βάση συνένεσης και εκμεταλλευόμενη τα θετικά της επιχείρησης. Να προβλέπουμε τι εξελίξει. Να προειδοποιούμε να ενεργούμε έγκαιρα, να αποφεύγουμε τα αρνητικά, που δεν είναι πάντοτε εφικτό, αλλά πολλές φορές γίνεται. Ξέρουμε την αγορά ή κάποια κομμάτια της. Οπότε έτσι ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους, τα αρνητικά. Και έτσι να συνεχίζει να υπάρχει επιχείρηση, η δραστηριότητα, η απασχόληση. Διαχείριση δίκαιη, ευφύη να μην γίνεται αυταρχικά, άδικα η αναδιάρθρωση. Να δικαιολογούμε γιατί την κάνουμε. Και όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι να έχουν ισότητα. Είδατε την Αρσελόρ; τι είναι την General Motors. Η μία περιφέρεια είναι αντιμέτωπη με άλλη. Ο ένας εργαζόμενος με τον άλλο εμείς να φροντίζουμε όλοι να βγαίνουν κερδισμένοι όλες οι επιχειρήσεις, να εμπλέκονται όλοι οι κοινωνικοί Γιατί έχουμε εδώ φαινόμενο το οποίο αφορά όλη την κοινωνία. Είναι κάτι που έχει πάρα πολύ σημαντικές επιπτώσεις στις βιομηχανικές περιοχές. Μιλούμε για εκατοντάδες χιλιάδων εργαζομένους δεν είναι ισόρο, ισο, ισομερός κατανοημένη. είναι συγκεντρωμένη σε αυτές τις περιοχές. Άρα, προσοχή για τις καταστροφικές συνέπειες στην οικονομία και στον άνθρωπο. Υπάρχει, υπάρχουν, υπάρχει τεκμήρια στο πόσο βλάπτεται η ανθρώπινη υγεία από τέτοιες ε, αποτυχίες. Θα πρέπει να είναι επικοδομητική αυτή η διαδικασία, υπάρχει εποπτεία και όλα αυτά θα θίξουν και θα βαρύνουν τα, τα αρπακτικά και όχι τις σωστές επιχειρήσεις. Με υπεύθυνο τρόπο επομένω θα περιορίσουμε τους κινδύνους. Να βγάζουμε μόνο τα θετικά. Όλες οι εταιρείε και δημοσίου συμφέροντος εταιρείε. Επίση, αυτοί που βγαίνουν χαμένοι από τι αναδιαρθρώσει θα πρέπει να βοηθούνται. Η Ευρώπη δεν υπάρχει για να παρέχει συμβουλέ. Η Ευρώπη υπάρχει για να βοηθά. Να βοηθά αυτού που βγαίνουν χαμένοι. Πάντα βγαίνουν κάποιοι χαμένοι και κάποιοι κερδισμένοι. Να είμαστε στο πλευρό του. Να του ανακυκλώσουμε. Του δίνουμε νέε ευκαιρίε. φορές τεχνολογική μεταβολή ε, και αυτή έχει αρκετέ επιπτώσεις και, αυτό να βοηθούμε. Το πνεύμα και η φιλοσοφία μας είναι ο κοινωνικό διάλογος. Διαβούλευση με τους εργαζομένου. Να δούμε επίσης πού είχαμε πιο μεγάλες επιτυχίες. σε ποιες χώρες. Ευελιξία και ασφάλεια ταυτόχρονα. Αυτή που σεβάστηκαν όχι μόνο την αλλαγή και την καινοτομία, αλλά και το διάλογο και τη δημοκρατία. Δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι το, η μοναδική μέρη είναι, είναι ο κύριος Μιτάλ να στο κάθε στο διαμέρισμα του στο Λονδίνο. Τι θα γίνει. Προσοχή και στις αγωγές από την Ασία θα πρέπει να χρειάζεται και, πάνω σε αυτό. Ε, διαβούλευση του εργαζομένου. Και έτσι οι υποχρεώσεις που έχουν να τηρούνται. Δεν είναι δυνατόν επιχειρήσεις μόνο να φροντίζουν για την αύξηση του κέρδους. Χρειάζεται κοινωνικό διάλογος. Αυτό το θέμα δεν είναι ιδεολογικό. Διαβάστε εδώ την επιστημονική τεκμηρίωση. Όλες οι επιτυχείς αναδιαρθρώσεις έγιναν με κοινωνικό διάλογο, με κοινωνική συνένεση και με την υποστήριξη των τοπικών περιφερειακών αρχών. Αυτή είναι η που θέλουμε να κάνουμε. Και θα την κάνουμε εάν έχουμε κατά νου πού θέλουμε να φτάσουμε, τι θέλουμε να πετύχουμε και να σταματήσουμε όλα να γίνονται στο βωμό της αγοράς και των μετόχων. Ο άνθρωπος είναι το πιο σημαντικό. Η αγορά πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και τι αποκεντρισμένε και οι ίδιε οι επιχειρήσει πρώτε-πρώτε. Και γι' αυτό, συνάδελφοι, ε, όπω είπα, πρόκειται τώρα να ξεκινήσει μια μεγάλη διαδρομή και να την κάνουμε χέρι-χέρι Πρόκειται εδώ πέρα για κάτι που δεν αφορά συγκεκριμένο κόμμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την Ευρώπη. Εμείς δεν μπορεί να είμαστε αδιάφοροι ε, στο, στο, στα προβλήματα, στις προκλήσεις, στις αλλαγές. Όμως εμείς μαζί να βοηθήσουμε όπου χρειάζεται και γι' αυτό και ελπίζω ότι να έχουμε πολλές τροπολογίες. Έχω ένα σωρό δίκτυα, με βοηθούν, πολλοί έχουν έρθει και με πλησίζουν να γίνει μια καλή έκθεση, μια έκθεση που να μην είναι δική μου. Μια έκθεση που να είναι οριζόντια. Όλοι μαζί να την κάνουμε εδώ στην Επιτροπή μας και αύριο ένα έκθεση όλου του Κοινοβουλίου. ιεραρχία και σωστή τάξη. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Λεμπή Φοντανιέ, δεδομένη τη σπουδαιότητα τη ομάδα τη. Η άλλη μου ζήτησε να παρεμβεί πρώτη και η ευγένεια ε, προς τις γυναίκες δίνει δυνατότητα από τις γυναίκες δίνει τη δυνατότητα στους φιλελεύθερου να μιλήσουν πρώτοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συγχαρητήρια για την έκθεση πρωτοβουλία του συναδέλφου μα, κυρίου Σερκά. Κανεί δεν μπορεί να έχει αντίρρηση ότι στη διαδικασία τη αναδιάρθρωση τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εμπλέκονται και να ενημερώνονται έγκαιρα. Έχουμε κοινό στόχο. Θέλουμε οι αναδιαρθρώσει να προκαλούν όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα, με όσο το δυνατόν λιγότερε απολύσει. Ω παρενέργειε θα πρέπει να είναι διαφανεί οι διαδικασίε προσχεδιασμένε και να εκτελούνται με τρόπο φιλικό προ του υπαλλήλου και προ του υπόλοιπου ενδιαφερομένους τη τοπική κοινότητα, ώστε να αποφεύγονται εκτενή κοινωνικά κόστη ωστόσο ως φιλελεύθεροι θα εξετάσουμε προσεκτικά τις λεπτομέρειες αυτής της έκθεσης και θα φροντίσουμε εν τέλει να μην αποτελεί βάρος για τις επιχειρήσεις που ήδη ε, ε, διέρχονται από μια διαδικασία που κοστίζει πολλά και δύσκολη. Επιθυμούμε να έχουμε ένα υγιές και υποστηρικτικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ η κυρία Λούπη Φοντανιά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον κύριο Σίγητη. Το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Βλέπω ότι έχει πολύ ισχυρέ πεπιθήσει. Ε, είναι μεγάλο το στίχημα αυτό και θα πρέπει όλοι να υποστηρίξουμε αυτή την έκθεση, η οποία σίγουρα είναι ενδιαφέρουσα και σημαντική. Επαναλαμβάνω, η συζήτησή μας αυτή είναι σημαντική για την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας. Υπόθηκε καθαρά από τον Αλεχάνδρο Σέρκας. Είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, χρειάζονται ανάκαμψη να επιστρέψουν στην ανάπτυξη ε, τηρώντας την επικουρικότητα σε όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά η κατάσταση δεν είναι αυτή που ήταν πριν από ένα χρόνο όταν και τότε μιλούσαμε για αναδιαρθρώσεις. Όσον αφορά την ομάδα μου είναι πολύ σημαντικό και για μένα προσωπικά να επιστήσουμε όλοι μας την προσοχή σε αυτά τα σημεία. Δηλαδή την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την πρόβλεψη όπως είπε ο Αλεχάνδρο όσον αφορά τις επιχειρήσεις μας. Καθημερινά ακούμε αναδιορθώσεις ξαφνικές. Είναι σημαντικό λοιπόν να αποφύγουμε τις εξωχωρήσεις αναθέσεις δραστηριοτήτων, ένα σημαντικό φαινόμενο που ε, λαμβάνει η χώρα εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρώπη. Ε, επιδεινώνεται όλο και περισσότερο σε όλες τις χώρες η κρατικοί μηχανισμοί θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή εργαλεία για να αποφεύγουν την διαφυγή επιχειρήσεων από τα κράτη-μέλη μα. Αλλά δύο σημεία που θεωρώ σημαντικά όσον αφορά το θέμα των αναδιορθώσεων είναι ότι πρέπει να ορίσουμε σαφώς τι θεωρούμε ότι είναι η αναδιάρθρωση, διότι ενδεχομένω ο ορισμός της αναδιάρθρωσης δεν είναι ίδιος σε όλες τις χώρες. Σκόπιμο θα ήταν λοιπόν να έχουμε έναν κοινό ορισμό. Ένα άλλο θέμα που θεωρώ θεμελιώδη σημασία ε, είναι η αρχή τη επικουρικότητα. Πρέπει να τηρούμε και να επακούμε στην ισχύουσα νομοθεσία στην εκαστοτέ χώρα. Καλό θα ήταν λοιπόν υπήρχε ένα βασικό σύνολο κανονισμών που θα ισχύει στα κράτη-μέλη εκεί όπου δεν υπάρχει νομοθεσία αυτού του τύπου. Και αυτό θα πρέπει να το μελετήσουμε, συμφωνώ. Επίση δεν πρέπει να ξεχνάμε να προσέξουμε ιδιαίτερα τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Άλλα σημεία στα οποία αναφέρεται η έκθεση είναι η κατάρτιση των εργαζομένων. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη να επιμείνουμε στην κατάρτιση των εργαζομένων αφού υπάρχει ήδη νομοθεσία σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων όσον αφορά την κατάρτιση. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό τόσο και η παρουσίαση όσο και η ουσία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια ισορροπημένη άποψη ώστε να διευκολύνουμε μια συμφωνία για την αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας. Θα πρέπει να είμαστε λογικοί όταν βρίσκουμε σημεία κοινά. Μιλάμε για δύο σημαντικές κατευθύνσεις αυτή που είναι υπέρ μιας ευρωπαϊκής οδηγίας και οι άλλοι που θέλουν να ακολουθήσουν έναν άλλο δρόμο πιο συγκεκριμένο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να το συζητήσουμε τόσο στο πλαίσιο της δικής μας επιτροπής μεταξύ των διαφορών ομάδων, αλλά είμαι και πεπισμένη ότι θα καταφέρουμε να επιτύχουμε μια συμφωνία και είμαστε έτοιμοι σε αυτές τι εποχές τόσο σοβαρή κρίση με τόσες καταστροφές για τόσους πολλού εργαζομένου. είμαστε έτοιμοι όπως είπε ο κ. Σίγητης, να αποφύγουμε την αποτυχία αυτής εδώ της έκθεσης εκ μέρους του ΕΛΚ. Λοιπόν, θεωρώ ότι σίγουρα θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Σιγητή, ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μεταξύ όλων μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριο Στομασμάνη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Βέβαια η συνάδελφος Στάινμπρουκ ευχαρίστως ε, ε, μας παρασύρει αλλά θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σέρκας για την έκθεση η οποία πολύ σωστά είπε ότι πρέπει να έχουμε μία έκθεση χωρίς ιδεολογία υπάρχει ιδεολογία αγοράς υπάρχουν αρχές τις οποίες πρέπει να εφαρμόζουμε διότι δεν είναι δυνατόν να κάνουμε κάτι διαφορετικό οι άνθρωποι χρειάζονται μία ρεαλιστική πολιτική σαφή η οποία μας ανοίγει δρόμους. Και όπως το είπες και εσύ όσον αφορά την Όπελ δεν είναι δυνατόν τα σημεία όπου υπάρχουν ε, ε, ορισμένα εργοστάσια να θεωρούνται σαν σημείο ενάρξεως μία διενέξεως για μεταφορά προς την Έση ή κάπου αλλού. Ε, πρέπει να υπάρξουν αποτελέσματα τα οποία θα επιτρέψει στους αρμοδιότητες διούς να λύνουν τα προβλήματα. Τι επιτύχαμε μέχρι στιγμής. Να υπάρχει μία εξασφάλιση εργασίας ε, για σειρά ετών αλλά χωρίς αυξήσεις μισθών η οποία είναι μία ε, ε, επιτυχία αλλά επώδυνη και κοιτάζουμε να διατηρήσουμε θέσεις στην Ευρώπη όχι μόνο μέσα στην Ευρώπη αλλά να διατηρήσουμε και τις θέσεις εκεί που υπάρχουν εκτός Ευρώπη Ευρώπης και να υπάρχουν εισαγωγές. Η ποιότητα, η αξιοπιστία αγορών σαν την Ισπανία, σαν τη Γερμανία μας δείχνουν ότι έχουμε μεγάλο παραγωγικό δυναμικό, παράγουμε ποιότητα, ελπίζουμε ότι το εκτιμούν οι καταναλωτές και δεν πρέπει να λέγουν ότι εφόσον ε, ε, το προϊόν αυτό απέτυχε προσπαθούμε να το χρηματοδοτήσουμε και πετάμε χρήματα. Δεν θέλουμε τέτοια και γι' αυτό είναι σημαντικό να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας. Επίσης μίλησα και με άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όχι μόνο την Όπελ και αυτές μου είπαν ότι όντως ε, έχουμε πολιτικές σε διάφορα σημεία της Ευρώπης και πρέπει καταρχήν να ξέρουμε ε, ποιο θα είναι το μέλλον, πώς θα διαγραφεί το μέλλον κατά τρόπον ώστε οι εργαζόμενοι να δουλεύουν λογικά να ε, προσφέρουν επαρκή ποιότητα και να ξεπερνάμε τα προβλήματά μας και γι' αυτό χαίρομαι ε, που θα γίνει αυτή η ακρόαση διότι είναι το, η κατάλληλη στιγμή για να μπορέσει να προχωρήσει και ελπίζουμε ότι η έκθεση αυτή θα στηριχθεί από καλές τροπολογίες για να προωθήσει το έργο της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα τον Αλεχάνδρο και ακούγοντας τον σχημάτισα την εντύπωση ότι ότι βρισκόμουν σε μια μεγάλη συνδικαλιστική διαδήλωση. Τόσο ενθουσιώδης ήταν με την παρουσίασή του. Δεν έχω να πω κάτι επί της ουσίας. Συμφωνώ γενικά με τα όσα προτείνει. Ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ωστόσο σε ορισμένα σημεία. Ο Αλεχάνδρο λέει ότι ότι χρειάζεται μακροχρόνια προετοιμασία ισχυρή ότι πρέπει να ετοιμαστούμε για τις μεταλλαγές, ότι πρέπει να προβλέψουμε πραγματικά τη διαδικασία, το πώς θα εξελιχθεί, ότι πρέπει να υλοποιήσουμε συστήματα κατάρτισης και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα κατά την άποψή μου είναι ότι ο κόσμος επιταχύνει όλο και περισσότερο. Σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε παγκόσμιες προκλήσεις και δεν έχουμε πλέον το χρόνο. Δεν προλαβαίνουμε να θέτουμε ερωτήματα Μπορούμε δηλαδή να αποφασίσουμε μονομερώς, μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι ε, αναγκαστικά, κάποιες λύσεις. Ε, σίγουρα μπορούμε αναγκαστικά και μονομερώς να επιβάλλουμε κάποιες λύσεις, αλλά αξίζει τον κόπο να κάνουμε κάτι τέτοιο. Θα μας επιτρέψει αυτό να προβούμε σε μεταλλαγές, αναδιαρθρώσεις κατάλληλες. Θα είμαστε βέβαιοι ότι αυτό θα διασφαλίζει απασχόληση για απολυμμένους θέτω αυτό το ερώτημα και γνωρίζω την απάντηση βέβαια. Η απάντηση κατά την άποψή μου είναι ότι όχι, δεν αξίζει τον κόπο να ακολουθήσουμε αυτή την οδό. Πράγματι είναι προτιμότερο να υλοποιήσουμε κείμενα που αφορούν το δικαίωμα για την κατάρτιση. Χρειάζομαστε επίση νομοθεσία ώστε να γνωρίζουμε πώς να διαχειριζόμαστε μία οικονομία σε πλήρη μεταμόρφωση. Και θα χρειαζόμαστε λύσεις κατάλληλες για όλους τους ενδιαφερομένους. Επ' αυτού μπορούν να επωφεληθούν όλοι οι αρχές, οι μισθωτοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Ίσως θα έπρεπε να παρακολουθούμε τις πληροφορίες, να έχουμε ε, τράπεζες ε, δεδομένων, ε, πιο εύκολες στη χρήση, πιο ευέλικτες. Συμφωνώ και με την ιδέα του το να έχουμε ένα καλό σχέδιο σε κοινωνικό επίπεδο μπορεί να βοηθήσει να καταλήξουμε σε καλές ή τουλάχιστον σε καλύτερες λύσεις. Επιτρέπει επίση τη διασφάλιση της ευελιξίας. Σε περι... Αν μειώσουμε την ταχύτητα των μεταλλαγών, οι επιχειρήσεις μπορεί να έχουν άσχημη αντίδραση και να δεσμευτούν σε λύσεις μη επιθυμητές. Και ίσως τελικά καταλήξουν οι επιχειρήσεις να μην εφαρμόζουν το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης και να επιλέξουν λύσεις ουσιαστικά επίθεσης προς τους εργαζομένους. Δεδομένων αυτών βρισκόμαστε υπό πίεση. Υπάρχουν ελάχιστες διαθέσιμες λύσεις. Θα το σκεφτώ εγώ ίδιος και δεσμεύομαι μαζί με την πολιτική μου ομάδα να προβληματιστούμε ώστε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε ρεαλιστικές λύσεις και πώς θα μπορούσαμε να εξετάσουμε όχι μόνο τις γενικές αρχές, αλλά και γεγονότα που ήδη έχουν λάβει χώρα και τα επερχόμενα γεγονότα, τα οποία δεν προλαβαίνουμε λόγω της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται ο κόσμος. Υπάρχουν άλλες ε, ομιλίες, ε, ομιλητές. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω τον συνάδελφο και φίλο κύριο Σέρκας για την, του, για την πρότασή του είναι μετρημένη και μας την παρουσίασε με τον συνδικαλιστικό ενθουσιασμό που γνωρίζουμε όλοι. Επί της ουσίας όμως είναι πολύ ισορροπημένη και προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα που βιώνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν πρώτα ο τρόπος ε, με τον οποίο σκέφτηκε ο κ. Τομασμάν... Πρέπει να προχωρήσουμε έχοντας υπόψη μας τι είναι η κοινωνική οικονομία της αγοράς. Υπάρχει χώρος για μια τέτοια πρωτοβουλία αφενός. Αφετέρου, αν θα μπορούσαμε σε ευρωπαϊκή κλίμακα να επωφεληθούμε, η Γερμανία συχνά καταδεικνύει άλλους με το δάκτυλο. Όλοι βέβαια έχουμε να μάθουμε πράγματα όσον αφορά τον κοινωνικό διάλογο και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων από τη Γερμανία. Ε, αν μπορούσατε να εξάγετε αντί σε αυτή την ποιότητα διαλόγου θα προσφέρετε τεράστια προσθέμενη αξία. Έχοντας αυτό λοιπόν υπόψη μας μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα διότι δεν ξεκίνησαν αυτή την πρωτοβουλία οι συντονιστές. Ήταν μάλλον εθελοντικοί τότε δεν είχαμε ακόμη προβλέψει σε ποιο βαθμό θα ε, τέριαζε με την πραγματικότητα που βιώνουν πολλές επιχειρήσεις σήμερα. Είδα πάλι αριθμούς χθε ε, στις εφημερίδες, ε, είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει. Φανταζόμαι λοιπόν, μπορώ να φανταστώ εύκολα, ότι θα κινητοποιηθούμε πολύ έντονα, ορισμένοι δηλαδή μάλλον φορείς θα κινητοποιηθούν έντονα για αυτή την έκθεση του κυρίου Σέρκας, δεν ξέρω αν είναι παρόντες εδώ στην αίθουσα, αλλά θα κάνουν ό,τι μπορούν για να εμποδίσουν μια τέτοια πρωτοβουλία. Εγώ πιστεύω ότι ως νομοθέτες, ε, δεδομένου του όσων έχουμε πει σήμερα και όταν όσων λέμε καθημερινά, θα ήταν κρίμα να τους ακούσουμε. Αν θεωρούμε ότι υπάρχει ένα ανθρώπινο κεφάλαιο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι αυτό είναι το κυριότερο μας ατού, θα πρέπει να βρεθούμε σε μια τέτοια θέση ώστε να μπορέσουμε να το ικανοποιήσουμε και να το αξιοποιήσουμε και να το αναδείξουμε περισσότερο από τη σήμερα. Τώρα το επιχείρημα της επικουρικότητας. Αυτό το επιχείρημα ακριβώς χρησιμοποιείται από όσους ε, κατά κάποιον τρόπο αντιτίθενται ε, στα ευρωπαϊκά ιδεώδη για να τα καταστρέψουν καλύτερα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο οι Ευρωπαίοι σε τι θα είχαν συμφέρον να εγκαταλείψουν τις χώρες που θα έλεγα εμβληματικές. Ε, η οικονομία που πάντα αναδεικνύεται ως παράδειγμα η γερμανική οικονομία ήταν μια οικονομία η οποία ήταν ικανή να διατηρήσει τη δημιουργία αξιών μέσω της βιομηχανικής παραγωγής. Με αυτό το πνεύμα πρέπει να ξαναβρούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να το ξαναβρούμε αυτό το πνεύμα χρειαζόμαστε νομοθεσία σε θέματα αναδιάρθρωσης διότι διαφορετικά αφήνουμε όσους συμπεριφέρονται όχι ως αφεντικά, ως βιομηχανία, αλλά ως διαχειριστές κερδοφόρων κεφαλαίων, κερδοσκοπικών κεφαλαίων, τους αφήνουμε να βελτιστοποιούν τα κέρδη τους ε, και να πηγαίνουν να επενδύουν αλλού, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω λοιπόν εγώ ότι υπό το κοινωνικό πρίσμα μπορούμε να έχουμε ένα φαινόμενο μόχλευσης ε, πολλαπλασιασμού για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, τηρώντας φυσικά την επικουρικότητα, αλλά αν σταθούμε μόνο σε αυτό το επιχείρημα, τότε θα παίξουμε το παιχνίδι όσων θέλουν το δικό τους μικρό μονοπόλιο και που θέλουν να λυλατήσουν το, ευρωπαϊκό, το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτώντα τι ε, πιο συγκεκριμένε προτάσει του Χάνδρο Σέρκα, κυρίω όσον αφορά την ενημέρωση και τη διαβούλευση με του εργαζομένου, υπάρχει μια συγκεκριμένη διάσταση για τι αναδιαρθρώσει. Διότι είδαμε πολλά κείμενα για την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων. Όταν εφηβήθηκε το τελευταίο κείμενο, στο τέλο, τη στιγμή τη ψηφοφορία, εγώ με τη δική μου πολιτική οικογένεια είπαμε, όχι αυτό δεν είναι εντάξει, δεν είναι αρκετό. Και ένας από τους λόγους που πραγματικά υπήρχαν ελλείψεις ήταν ο τομέας των αδιαρθρώσεων. Ίσως αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε όλο το φάκελο για την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων, αλλά ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την πρωτοβουλία για να στοχεύσουμε ακριβώς αυτό τον τομέα και τις ελλείψεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτές είναι κάποιες προτάσεις που ήθελα να κάνω. Χαίρομαι ιδιαίτερα, ιδιαίτερα ικανοποιημένη από αυτή την επικοδομητική συζήτηση. Κύριε Σίγητα, έχετε το λόγο για να ολοκληρώσετε. Θα μου επιτρέψουν οι συνάδελφοι να αρχίσω με κάτι το συμπαθητικό, το γενικό ότι εγώ αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι ο συνδικαλισμός. Ο συνδικαλισμός άλλωστε είναι κάτι πάρα πολύ πάρα πάρα πολύ ευάλωτο ευαίσθητο λεπτό είναι ότι πρόκειται για αγώνα που έχω δώσει μια ζωή. Νομίζω ότι στη σημερινή συγκυρία στην Ευρώπη Είμαστε στριμωγμένοι εμείς οι πολιτικοί, στριμωγμένοι και καλούμεθα να δώσουμε λύσεις και όχι λόγια. Και θα είχα αποτύχει εάν δεν τολμούσα να μπω στην αρένα, να αντιμετωπίσω το πρόβλημα και να κάνω κάτι που θα είναι βασισμένο όχι σε ιδεολογήματα, αλλά σε κάτι πάρα πολύ πρακτικό όπως η Αρσελόρ, η Όπελ όλα αυτά τα οποία αφορούν ανθρώπους, γυναίκες, άντρες, χωριά, πόλεις, που είναι μόνοι όλοι αυτοί που κινδυνεύουν, αισθάνονται μόνοι και δεν θέλω να τους αγνοούμε. Εντάξει, φανατισμό νιώθω, ας πούμε πάθος και, και φανατισμό, πούμε για το ποδόσφαιρο, για άλλα πράγματα. Αλλά, Τόμας, αυτό το οποίο θέλω είναι να γίνεται αναδιάρθρωση ευφυής. Δεν είναι θέμα δεξιάς αριστεράς. Θέλω να βγαίνουν όλοι κερδισμένοι. Οι εργαζόμενοι και ταυτόχρονα και οι επιχειρήσεις. Τι έγινε στην ε, Θαραγώθα. Εκεί είχαμε διάλογο, είχαμε συνεννόηση. Χιλιάδες θέσεων εργασίας σωθήκανε και μέσα σε τρεις εβδομάδες εκεί στη Φιρουέλα, στη Θαραγώθα, κατάφεραν έτσι να, να το σώσουν. Ενώ αλλού, αλλού έκλεισε η επιχείρηση εκεί κοντά στην ίδια πόλη. Γιατί δεν υπήρχε υπευθυνότητα. Για... Το μόνο που του ενδιαφέρει είναι να παίζουν με τι μετοχέ στα χρηματιστήρια. Να, με τι φανατίζομαι. Να, τι θέλω. Θέλω διακαώς να συμφωνήσουμε. Θέλω να λύσουμε τα προβλήματα και είμαι ανοιχτό και ήδη πάρα πολύ έχουμε ασχοληθεί με αυτό το κείμενο και θα κάτσω εγώ και θα συζητήσω με του οικειοδησηγητέ, θα τα συζητήσουμε όλα. Και η μόνη μου κόκκινη γραμμή θα είναι ότι τα, τα πράγματα δεν μπορούν να συγχυστούν όπω είναι τώρα. Γιατί όπω είναι τώρα τα πράγματα, είναι το, το, αυτό το 10% που χάσαμε από τη βιομηχανική μα ισχύ. Δεν είναι δυνατόν να παρατηθούμε και να ε, θεωρήσουμε ότι θα πάει να γίνει έρημο βιομηχανική Ευρώπη. Πάνε τα, τα ταμεία, οι συντάξει, όλα. Άμα κλείνουνε τα εργοστάσια χωρίς κανείς να σκέφτεται τον άνθρωπο. Όλους αυτούς που υφίσταται τις συνέπειες επομένως. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Ο διάλογος θα είναι επικοδομητικός. Ναι, θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Δεσμεύομαι γι' αυτό. Ο φίλος Σαβαρή βεβαίως και θα βρει ανταπόκριση σε όλες αυτές τις προστάσεις. Πρακτικά πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, ε, θα μπορέσουν να κατατεθούν σε λογικά περιθώρια οι τροπολογίες μέχρι τις 9 Ιουλίου το μεσημέρι για να τις ε, εξετάσουμε στις 17-18 Σεπτεμβρίου και ε, να ψηφίσουμε στην Επιτροπή 8-9 Οκτωβρίου και ε, αν είναι δυνατόν να περάσει την πρώτη Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Ε, ερχόμαστε τώρα στο σημείο 17 της ημερησίας διάταξης και δίνω το λόγο στην κυρία Ρουντζόλη για την γνωμοδότησή της σχετικά που απευθύνεται προς την ΙΜΚΟ για την τροποποίηση των επαγγελματικών προσόντων σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Κυρία Ροντσούλη, έχετε το λόγο. Λοιπόν, η τρέχουσα οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, η 2536, έφερε ένα δίπλο πλεονέκτημα τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τις επιχειρήσεις. Ευνόησε την κινητικότητα ειδικευμένων εργαζομένων και συνέβαλε στην ανάπτυξη διασυνοριακών υπηρεσιών. Η αφαίρεση ορισμένων εμποδίων της κινητικότητας τόνωσε την ανταγωνιστικότητα και δημιούργησε νέες θέσεις απασχόλησης. Ωστόσο, το ποσοστό κινητικότητα επαγγελματιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακόμα χαμηλό. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, μόνο το 28% των πολιτών εξετάζει, αξιοποιεί τη δυνατότητα μεταφοράς στο εξωτερικό για το επαγγελματίο του και φυσικά πάντα λόγω των δυσκολιών που σχετίζονται με τα επαγγελματικά προσόντα. Η κινητικότητα, όπως γνωρίζουμε, βοηθά σε αύξηση των ικανοτήτων και γνώσεων μεταξύ κρατών μελών, που μπορεί επίση να βελτιωθεί μέσω μια κοινή προσέγγιση, ώστε να διασφαλίζει υψηλή ποιότητα ε, κατάρτισης και εκπαίδευση. Η αγορά των επαγγελματών ε, αναβαθμίζεται συνεχώ και εξελίσσεται συνεχώς παραδοσιακά επαγγέλματα ε, δίνουν τη θέση τους σε νέα πιο ειδικευμένα επαγγέλματα. Το σημερινό σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων απαιτεί αναβάθμιση για μεγαλύτερη ευελιξία, αναγνώριση των ικανοτήτων και μείωση του διοικητικού κόστους. Η Επιτροπή λοιπόν προτείνει αναθεώρηση για την επαναδρομολόγηση της εσωτερικής αγοράς, την πρόσφορα νέων ευκαιριών επαγγελματικών και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των κρατών μελών όπου υπάρχει έλλειψη ε, ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Τα καινοτόμα στοιχεία αυτή της πρόταση είναι πολλαπλά. Το πιο σημαντικό είναι το επαγγελματικό, το ευρωπαϊκό επαγγελματικό δελτίο, επαγγελματικό διαβατήριο δηλαδή. Η Κομισιόν προτείνει ένα νέο επαγγελματικό διαβατήριο που θα βοηθά σε πιο απλή αναγνώριση των προσόντων καθώς και μείωση του διοικητικού κόστους ε, για την αναγνώριση των διαφόρων διπλωμάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επενθυμίζω, 15 Νοεμβρίου του περασμένου έτους σε μια έκθεση για την επαναδρομολόγηση της εσωτερικής αγοράς ψήφισε θετικά ένα ψήφισμα όπου υπογραμμίζεται ότι ένα εθελοντικό επαγγελματικό διαβατήριο θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για να διευκολύνει την κινητικότητα σε ορισμένα επαγγέλματα. Η Κομισιόν, Επιτροπή προτείνει αυτό το διαβατήριο σε εθελοντική βάση, αφήνοντας την ελευθερία στα κρατημέλη να επιλέξουν τον οργανισμό που θα το εκδίδει. Η άποψή μου για αυτό το ευρωπαϊκό διαβατήριο είναι να γίνει υποχρεωτικό. Μετά από μια μελέτη αντικτύπου που ολοκληρώθηκε για τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου διαβατηρίου και αξιολογώντας φυσικά τα κόστη και τους χρόνους φυσικά. Μάλιστα πιστεύω ότι η υποχρεωτική υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού διαβατηρίου σε σύγκριση με το εθελοντικό μιλάμε εδώ για ένα εργαλείο Εάν είναι θελοντικό, τα κράτη-μέλη έχουν τάση να μην υιοθετούν τέτοιου είδους διαβατήρια. Το επαγγελματικό διαβατήριο, το ευρωπαϊκό, θα μειώσει τα κόστη που υποχρεούνται να ε, καταβάλουν ε, οι επαγγελματίες για την αναγνώριση των διπλωμάτων ή της ισοτιμίας τους. Σήμερα ένας νοσοκόμος για να αναγνωριστεί το πτυχίο του ξοδεύει 140 ευρώ στην Αυστρία, 200 στην Ιρλανδία στην Ουγγαρία και 300 στην Φιλανδία. Ένας μηχανικός από 200 στην Αυστρία και την Πολωνία και ένας ε, θεραπευτής, για παράδειγμα στην Ολλανδία, 600. Όπως βλέπουμε υπάρχει τεράστια διαφοροποίηση η νέα διαδικασία, προβλέπει επίσης τον στόχο απλούστευσης και επιτάκυνσης της διαδικασίας αναγνώρισης. Εγώ πρότεινα τέσσερις εβδομάδες. Αντίθετα από την Κομισιόν που προτείνει μόλις δύο. Ωστόσο αυτό μου φαίνεται πολύ μικροχρονικό διάστημα, δύο εβδομάδες. Επιπλέον η πρότασή μου είναι να γίνει πιο διαφανής η διαδικασία. Προτείνω να εξαλείψουμε από την πρόταση της Κομισιόν την σιωπηρή ε, συμφωνία. Λέει η Κομισιόν δηλαδή στην πρότασή της ότι μετά από δύο εβδομάδες έχει κανείς δικαίωμα στο Ευρωπαϊκό Διαβατήριο εφόσον δεν ε, υπάρχει σιωπηρή συμφωνία. Αλλά δεδομένης τεράστιας γραφειοκρατίας που υπάρχει σίγουρα θα χρειαστεί μια σιωπηρή συνένεση. Αλλά μια σιωπηρή συνένεση εδώ πέρα δεν καθιστά διαφανή ε, τη διαδικασία αυτή του Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου το κάθε αίτημα θα καταγράφεται στο πληροφορικό σύστημα της εσωτερικής αγοράς. Στα κράτη-μέλη εκχωρείται απόλυτη ελευθερία επιλογής των κριτηρίων βάσει των οποίων θα καθορίζουν τα επαγγέλματα για τα οποία θα προβλέπεται κατά προτεραιότητα έκδοση του επαγγελματικού διαβατηρίου. Κατά Στη γνωμοδότησή μου προτείνω όσον αφορά την νέα προτεραιότητα έκδοση τουλάχιστον να κάνουμε διάκριση των κριτηρίων, δηλαδή το επάγγελμα να ρυθμίζεται τουλάχιστον από πέντε κρατημέλη, να έχει υψηλέ δυνατότητες κινητικότητας όπως οι νοσοκόμοι και να παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες και για τις ενώσεις της κατηγορίας. Αντιθέτως όσον αφορά την ε, έκδοση χωρίς προτεραιότητα το διαβατήριο θα προτείνεται σε επαγγέλματα νομικώς κατοχυρωμένα, αρχιτέκτονες, μηχανικούς και το καθώς και σε μη νομικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα όπω για παράδειγμα οι ταξιδιωτικοί οδηγοί δεν αναγνωρίζονται ως επάγγελμα σε όλα τα κράτη-μέλη. Ένα άλλο βασικό σημείο είναι η μερική πρόσβαση στο επάγγελμα. Βασισμένη στην ομολογία του δικαστηρίου, η Κομισιόν προτείνει να εισάγουμε στην οδηγία την έννοια της εν μέρη πρόσβασης. Της μερικής πρόσβασης αυτό το εργαλείο θα μπορούσε να διασφαλίσει νομική βεβαιότητα για τους επαγγελματίε, επειδή τους δίνει τη δυνατότητα να ασκούν το επάγγελμα χωρίς απαραίτητα να ολοκληρώνουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης για να ολοκληρώσουν την ήδη υπάρχουσα εκπαίδευσή του στα κράτη-μέλη μπορούν πάντα σύμφωνα με την Κομισιόν να αρνηθούν την μερική πρόσβαση εφόσον υπάρχει αιτιολογημένη ε, αιτιολογημένος λόγος γενικού ενδιαφέροντος ε, όπου επιβεβλημένος μόνος τέτοιος λόγος αφορά τη δημόσια υγεία κατά την άποψη της Κομισιόν κατά την έποψή μου τον αναφέρουμε μόνο τη δημόσια υγεία σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογής μόνο για συγκεκριμένα επαγγέλματα, δηλαδή όσους ας πούμε σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, γιατρούς, νοσοκόμους, παραϊτρικά επαγγέλματα και ούτω καθεξής. Πιστεύω λοιπόν, και το αναφέρω στην πρότασή μου, Επίσης και το δικαστήριο είχε αναγνωρίσει και άλλες ε, επιβεβλημένες αιτίες το να προσθέσουμε σε αυτή τη λίστα περισσότερες ε, ε, ώστε η άρνηση ε, μερικής ε, πρόσβασης να μπορεί να αφορά και άλλα επαγγέλματα, δηλαδή και άλλες επιβλημένες αιτίες θα μπορούσαν να είναι η δημοσία υγεία, η προστασία των καταναλωτών, η δημοσία τάξη, το σύστημα διατροφικής ασφάλειας, επισητιστικής ασφάλειας και άλλοι. Το άλλο σημείο αυτής της έκθεσης είναι οι ελάχιστες απαιτήσει κατάρτισης ε, εκπαίδευσης. Ο εξυγχρονισμός της τρέχουσας νομοθεσίας ε, βασίζεται στις ελάχιστες απαιτήσει εκπαίδευσης ώστε να παρακολουθούμε τα προγράμματα τα εκπαιδευτικά για το κάθε επάγγελμα. Αυτό το σημείο το οποίο είναι ιδιαίτερα επίμαχο αφορά κυρίως τους τομείς των νοσοκόμων και για τις ε, μαμές. Η Κομισιόν για τις ΜΕΕΣ 12 χρόνια κατάρτιση προβλέπεται για αυτού του είδους τα επαγγέλματα. Αυτό ισχύει ήδη σε 24 κράτη-μέλη. Για αυτό το σημείο συναντάμε ισχυρή αντίσταση κυρίως από τη Γερμανία. Τόμας, ε, αγαπητέ, και ε, λίγο από το Λουξεμβούργο, διότι στη Γερμανία και το Λουξεμβούργο υπάρχει κατάρτιση αντίστοιχα 10 και 11 ετών σε σχέση με τα 12 που προτείνει η Κομισιόν. Όσον αφορά εμένα, δική μου προσωπική μου άποψη, έχοντας ζήσει πολλά χρόνια σε νοσοκομείο πριν κάνω αυτή τη δουλειά, τα 12 χρόνια θα πρέπει να διατηρηθούν. Απλά για να σας ε, δώσω μια παραπάνω πληροφορία και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτών των επαγγελμάτων που συγκεντρώνει 34 εθνικές ενώσεις υποστηρίζει την πρόταση της Κομισιόν και μάλιστα ορισμένες γερμανικές ενώσεις την υποστηρίζουν. Ενώσεις αυτών των επαγγελμάτων υποστηρίζουν αυτά τα 12 χρόνια. Τι να κάνουμε υποστηρίζουν τα 12 χρόνια. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Πάντα όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις κατάρτισης, εκπαίδευσης τις επόμενες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ολοκληρώσει την τεχνική αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων του νοσηλευτικού προσωπικού που έχει εκπαιδευτεί σε Πολωνία και Ρουμανία, των οποίων οι που σπουδών ε, χορηγήθηκαν πριν το 2004, δηλαδή πριν από, την, πριν από την ένταξη των δύο αυτών κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η κατάρτιση φυσικά πριν το 2004 ήταν πολύ, χαμηλότερο πολύ χαμηλότερη, πολύ μικρότερη από δεκαέτη. Ένα άλλο σημείο αυτής της έκθεσης είναι τα αντισταθμιστικά μέτρα, τα μέτρα αποζημίωσης. Κάθε κρατος μέλος, εφόσον το θεωρεί απαραίτητο, μπορεί να εισαγάγει ε, αντισταθμιστικά μέτρα, επιπλέον εξετάσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Ωστόσο, εγώ προτείνω οι μηχανισμοί επαλήθευσης των ε, πρακτικών και θεωρητικών ικανοτήτων θα πρέπει να εγγυώνται το σεβασμό της διαφάνειας και της αμεροληψίας. Συνεπώς, δεν πρέπει να επιβαλούνται κριτική μεταχείριση. Επιπλέον, η τυχόν απόφαση εισαγωγής αντισταθμιστικού μέτρου. Ένα λεπτό δώστε μου έχω σχεδόν τελειώσει, θα πρέπει να αιτιολογείται λεπτομερώς. Ένα πρόβλημα φυσικά είναι η γλώσσα, ένα άλλο πρόβλημα αφορά του συμβολιογράφους που η Κομισιόν προτείνει να εισάγουμε πλήρως ε, σε αυτή την οδηγία και φυσικά τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν και εγώ απλά το αναφέρω. Επίσης υπάρχουν τα στάζ ε, με αμοιβή, εκπαιδευτικά προγράμματα με αμοιβή και τα κέντρα που θα γίνουν κέντρα υποστηρίξης και συμβουλευτικής υποστήριξης. Τέλειωσα, έκοψα πολλά. Απλά σας υπενθυμίζω ότι 10 Ιουλίου, 12 η ώρα το μεσημέρι, είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Ευχαριστούμε πολλά. Λοιπόν, ε, θα μπορούσαμε να σε ακούμε μία ώρα ακόμη, ευχαρίστως, αλλά ο χρόνος περνάει και έχουμε τώρα ε, τέσσερις ε, ομιλητές. Οπότε, για να είμαστε δίκαιοι, ο καθένας θα μιλήσει μόνο δύο λεπτά. Όχι παραπάνω, συμφωνείτε? Έχουμε ακόμη τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την γνωμοδότησή της και εγώ επεξεργάζομαι αυτό το θέμα στην Επιτροπή ΙΜΚΟ και θα σχολιάσω στα σύντομα διάφορα θέματα που έθιξε η συγγήτρηση. Καταρχήν όσον αφορά το επαγγελματικό δελτίο, την επαγγελματική κάρτα ε, και πιστεύω ότι δεν είναι εφικτό να είναι ε, εθελοντικό ή οικειοθελές και νομίζω ότι έχουν συμφωνήσει οι πολιτικές ομάδες ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μια εθελοντική κάρτα διότι δεν είναι τόσο εύκολο να ισχύσει αυτή η οικειοθελες και νομιζω οτι εχουν συμφωνησει πολιτικες ομαδες οτι Όσον αφορά τη μερική πρόσβαση, ε, ναι μεν αντιλαμβανόμαστε τις περιπτώσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαστηρίου αλλά τουλάχιστον στον τομέα της ε, υγειονομικής περίθαλψης είναι πολύ επιφυλακτική, πολύ. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μία σωστή ισορροπία. Όσον αφορά το χρόνο, διάφορα επαγγέλματα μας το έθιξαν ότι ε, δύο εβδομάδες δεν είναι δυνατόν και θα οδηγούσε σε απόρριψη της αναγνώρισης των προσόντων. Οπότε ίσως σωστά είπατε ότι χρειάζονται τέσσερις εβδομάδες και θα περιοριστώ σε αυτά τα σχόλια τώρα. Ωραία, η Μέρι Χάρκινγκ τώρα για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πρώτα πρώτα. Θέλω να πω κάτι για την Άντια που είναι ισχυώδης και δεν μπορούσε να παραστεί. Ευχαριστώ επίσης ε, την εισηγήτρια. Ε, είναι υπέρ ε, της υιοθέτησης αυτής της κάρτας του διαβατηρίου και συμφωνούμε για τις ευκαιρίες που δίνονται ο σκοπός είναι να εστιάσουμε την προσοχή μας στο να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία. Μέχρι τα 12 με αυτά είναι η γενική παιδεία, η βασική παιδεία, όσον αφορά το τομέα της υγείας, γιατί ακριβώς και οι νοσοκόμες και οι ΜΕΣ ε, είναι επαγγέλματα υψηλής ευθύνη. Και ε, να δούμε επίσης τι γίνεται και με τις ελλείψεις προσωπικού σε αυτές τις χώρες. Έχω δύο παρατηρήσεις, αφού ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία, δικές μου παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα για αυτό το επαγγελματικό διαβατήριο, την κάρτα, ε, καλή ιδέα. Όμως, προσοχή, όταν μιλάμε για τον τομέα της υγείας, κατά τη γνώμη μου, δεν αρκεί η απαρίθμηση των δεξιοτήτων. Γιατί πολλές φορές, ε, σε πολλά κρατημέρια στο δικό μου, είχαμε κάποιους που εργάζονται στον τομέα της να πρέπει να πάνε σε άλλη χώρα μέλος εκεί να χρειάζεται να έχουν αυτές τις πληροφορίες και να μην τις έχουν, μπορεί να το αποδείξουν τέλο πάντων. Οπότε είναι σωστό, ίσως αυτά να μπουν πάνω στην κάρτα. Κάτι άλλο τρόπο θα σας πω. Και... ότι όσον αφορά την κατάρτιση των γιατρών, έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα. Όταν κάποιος ήδη έχει σε κάποια σχετική επιστήμη δίπλωμα, μπορεί να γίνει γιατρός με τέσσερα χρονιά σπουδές, όπως γίνεται σε ΙΠΑ, Καναδά και Αυστραλία. Και αν ε, το προαπαιτούμενο της ε, πενταετίας επιβληθεί, θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Πάντως θα υποβάλω σχετικά τροπολογία. Ωραία. Αν μπορεί και ο επόμενος ε, λιγότερο από δύο λεπτά είπε σε ήδη ε, ποιο είναι το πρόβλημα στη Γερμανία και στην ε, Ουγγαρία παραδείγματος χάνει τα 10 χρόνια γίνονται 12 οπότε αποκλείονται πολύ οι ΜΕΕ στη Γερμανία όπου έχουμε πολύ καλή επαγγελματική κατάσταση αλλά έχουμε και ένα μεγάλο κενό και χρειάζεται μία κάλυψη. Είχαμε καλό πολύ καλό επίπεδο ε, ε, του ε, επαγγελματικού δυναμικού και υπάρχουν βέβαια άλλες χώρες που δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες και νομίζω ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Θα μπορούσε να υπάρξει μια συμβιβαστική λύση διότι όπως είπες υπάρχει μια διεθνής Ένωση, και μιλάμε για τουλάχιστον 10 χρόνια οπότε τότε μπορεί αυτά να συμβιβαστούν κάπως έτσι συμβιβαστικά και τα υπόλοιπα θα μας επιτρέψουν να τα κοιτάξουμε ε, ε, στη συνέχεια. Με τα χαρά σας λέω ότι ε, μίλησα λιγότερο από ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και θα πρέπει να προσέξουμε όσον αφορά την προσβασιμότητα. Δεν είναι θέμα ε, μόνο η παιδεία και η ιατρική, αλλά και αλλού και αλλού. Ας πούμε αυτοί που δουλεύουν ε, με γερανούς, ε, εξκαφείς και αυτά, ο, παντού, παντού, παντού, όπου υπάρχει κίνδυνος και χρειάζεται προηγουμένη κατάρτιση. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η κάρτα, αυτό το διαβατήριο με τις πληροσχετικές πληροφορίες. Επίσης, τελευταίο, θα πρέπει να δούμε ε, τι νόημα έχει να μείνουν να μείνουν γλωσσικοί περιορισμοί και κάποιος θα πρέπει να δουλεύει επομένως να δούμε ανάλογα τον τομέα τι θα γίνει. Τόμας. Αγαπητέ Όλε, νομίζω ότι όλα τα κατάφερε θαυμάσια. Ε, το ίδιο συμβαίνει και με το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι πάτε καλά. Λίντια, ξέρω ότι και εσύ ενδιαφέρεσαι για το ποδόσφαιρο. Οι Ιταλοί πάνε καλά και οι Ισπανοί και οι Γερμανοί. Οπότε εσύ έχεις ε, τον τελευταίο λόγο. Τους άκουσα όλους, δεν έχω να πω τίποτα. Έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε με τα επόμενα σημεία της ημερησίας διάταξης. Ευχαριστώ. Σας αναφέρω ότι η προθεσμία για τροπολογίες είναι 10 Ιουλίου 12 το μεσημέρι όπως είπε ήδη η Λίντια και τώρα μπορώ να δώσω το δικαίωμα στην Πρόεδρο να επανέλθει στην Προεδρία της. Hm. Λοιπόν, Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο Τόμας Μαν που μου επέτρεψε να επανέλθω στην Προεδρία για να σας πω το 18 και 19 δεν θα συζητηθούν σήμερα διότι δεν έχουμε πια χρόνο και άρα θα συζητηθούν αύριο ακριβώς μετά τις ψηφοφορίες και ευχαριστώ τους διερμηνείς και όλους τους συμμετέχοντες οι οποίοι παρέμειναν ως το τέλος και σας δίνω ραντεβού για αύριο. Καλό βράδυ.